Good morning, ladies and gentlemen. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Θα αρχίσουμε σε ένα λεπτό. Γι' αυτό παρακαλώ καθίστε. Και πάλι καλή σας μέρα. Και καλώς ήρθατε στη δεύτερη ημερίδα του σεμιναρίου μας που έχει να κάνει με τη δημιουργία ενός κοινού συστήματος ασύλου και δίκαιου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα αρχίσουμε με κάποιες ανακοινώσεις πρώτα για να έχουμε τελειώσει με τα πρακτικά. Το πρώτο είναι για σας που χρησιμοποιείτε Wi-Fi υπάρχουν νέοι κώδικες σήμερα. Αλλάζουν κάθε μέρα στο κοινοβούλιο. Θα τους βρείτε σε κάποια σημεία εδώ στην αίθουσα. Βλέπω ένα είναι εκεί δεξιά μου. Επίσης μπορείτε να υπογράψετε στον κατάλογο των παρόντων δεξιά πάντα. κάτω από την κενή καμπίνα διαρμηνίας. Για να συνοψίσουμε λοιπόν λίγο, τι κάναμε χτες. Χτες αρχίσαμε με το πρόγραμμα και είχαμε ανταλλαγή απόψεων με ευρωβουλευτές της Σεσίλια Πίλστρομ πρώτα απ' όλα, που είναι η συγγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη δημιουργία ακριβώς ε, αυτού του νέου συστήματος ασύλου. Στη συνέχεια είχαμε ανταλλαγή απόψεων με τους σκιώδεις εισηγητές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μετά είχαμε την Σόφη Μαγκένης από την ύπατη αρμοστία για τους πρόσφυγες του ΟΓΕ. Μετά Ακούσαμε τον Επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο. Σας θυμίζω ότι έχουμε διερμηνία, έτσι, οπότε να ξέρετε ότι όταν μιλάτε, όταν θέλετε να υποβάλλετε κάποια ερώτηση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μητρική σας γλώσσα. Αν είναι τα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά, τα ιταλικά, τα ελληνικά, τα ισπανικά, τα βουλγαρικά και τα ουγγρικά. Αυτέ είναι οι γλώσσες στις οποίες μπορείτε να υποβάλλετε τις ερωτήσεις σας. Τώρα, για το χρονοδιάγραμμα. Αρχίζουμε τώρα με τον κύριο ομιλητή μα και στη συνέχεια ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου θα έρθει στις 11 και 4, όχι 11 και 30, 11 και 4, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Συνεπώς πρέπει να γίνουν όλα νωρίτερα κατά ένα τέταρτο, που σημαίνει ότι δεν θα διακόψουμε για καφέ. Μπορείτε να πάρετε καφέ, αλλά δεν θα διακόψουμε. Στις 10 και 30 θα περάσουμε στο επόμενο πάνελ και στις 11 και 4, όπως σας είπαμε, 11 και 45 θα έχουμε τον πρόεδρο μαζί μας. Αν δεν έχουμε αρκετό χρόνο για τους προσκεκλημένους μας, μπορούμε μετά την συνάντηση με τον πρόεδρο να συνεχίσουμε. Θα προσπαθήσουμε. Θα δούμε πώς θα πάει. Συνεπώς, όταν υποβάλλετε ερωτήσεις, να λέτε πρώτα απ' όλα ποιος είσαστε, το όνομά σας, ποιον εκπροσωπείτε και για χάρη των διερμηνέων σας παρακαλώ να μην μιλάτε πολύ γρήγορα, λέει ο πρόεδρος. Χωρίς άλλη καθυστέρηση λοιπόν αρχίζουμε με το πρόγραμμά μας και καλωσορίζω εδώ τον κύριο Νταμιά Καρέμα που είναι ο δήμαρχος της Grand Ascent. Πρόκειται για μια πόλη που βρίσκεται στη Βόρεια Θάλασσα, στη Γαλλία. Είναι στη Μάνχη δηλαδή. Και επειδή μιλάμε για το άσυλο και την μετανάστευση, καταλαβαίνετε γιατί τον έχουμε μαζί μας. Στην Grand Saint υπάρχουν 21.000 κάτοικοι. Και τα τελευταία χρόνια είχαν να αντιμετωπίσουν πολλές και διαφορετικές καταστάσεις. Ο κύριος Καρέμ από το 2001 είναι δήμαρχος στην πόλη αυτή, 16 χρόνια δηλαδή. Οπότε έχει δει πολλά. Θα του δώσω λοιπόν το λόγο ευθύ αμέσω, ώστε να μοιραστεί μαζί μας τις εμπειρίες του και να μας πει τι ακριβώς έχει δει όλα αυτά τα χρόνια. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Καρέμ. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ για την πρόσκλησή μας σήμερα το πρωί. Σας καλημερίζω όλους. Θα σας διηγηθώ λίγο πολύ την ιστορία. Τι έγινε δηλαδή με την υποδοχή των προσφύγων στο δικό μου Δήμο, στη δικιά μου πόλη, που όπως είπε και ο συντονιστής μας εδώ, βρίσκεται στη Βόρεια Θάλασσα δίπλα στην Ντουκένκη λίγα χιλιόμετρα από το Καλέ. Είναι μια βιομηχανική πόλη, πρόσφατη, σχετικά από το 1960. Προηγουμένως ήταν μια μικρή πόλη αγροτική με 600 κατοίκους και φτάσαμε στις 25.000 που δουλεύουν στη βιομηχανία. Είχαμε την Ούζινορ μέχρι πρόσφατα που μετά έγινε Αρσελόρ και Αρσελόρ Μετάλ σήμερα. Για να δουλέψει κανείς το εργοστάσιο αυτό και για να χτιστεί το εργοστάσιο αυτό, το γαλλικό κράτος οργάνωσε το εξή. Πήγε και βρήκε εργάτες στην Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Αλγερία, το Μαρόκο, γιατί χρειαζόμαστε εργατικό δυναμικό στη χώρα μας τότε, μετά τον πόλεμο, καταλαβαίνετε, για να ενισχύσουμε την οικονομία μας. Και το θυμίζω αυτό, γιατί αυτό που συμβαίνει σήμερα με τους πρόσφυγες δεν είναι άσχετο με το τότε. Σήμερα Είμαστε σε βιομηχανική κρίση. 24% είναι η ανεργία στην πόλη μου. 33% των νοικοκυριών ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας και το ετήσιο μέσο εισόδημα είναι 9.600 ευρώ ανά νοικοκυριό. Σας τα λέω αυτά για να καταλάβετε ότι έχουμε να κάνουμε με μια φτωχή πόλη, με ένα πληθυσμό που αντιμετωπίζει σημαντικά κοινωνικά προβλήματα και τελικά όταν εξηγούμε τα της υποδοχής καταλαβαίνετε πώς ε, τα υποδέχονται όλα αυτά οι πολίτες. Όταν έκλεισε η Σανκάτ το 2002, κάποιοι πρόσφυγες ήρθαν κοντά στο κέντρο της πόλης, σε μια άδεια περιοχή, γιατί έχουμε ένα βενζινάδικο στο διαδρομή που πηγαίνει στο Καλέ και υπήρχαν διάφοροι οι οποίοι εκεί προσπαθούσαν να μπουν στα φορτηγά. Ερχόντουσαν, μέναν 24 ή 48 ώρες το πολύ και μετά φεύγανε. Διάφορες οργανώσεις ασχολήθηκαν για να τους προσφέρουν τροφή, ρούχα. Και αυτό έγινε από το 2002-2004 μέχρι το 2008 όπου ήρθαν οι διάφορες οργανώσεις, μας βρήκανε, είχε μείον 15 το 2008 το χειμώνα και για πρώτη φορά υπήρχαν και γυναίκες και παιδιά μεταξύ των προσφύγων αυτών. Οι οργανώσεις ε, λοιπόν ήταν ανήσυχε ότι θα πεθάνουν ε, τα παιδιά, οι γυναίκες από το κρύο. Οπότε ήρθαν σε επαφή μαζί μου και εγώ ζήτησα από τις υπηρεσίες μου να τους διαθέσουν μια θερμενόμενη σκηνή γιατί όποιο βρίσκεται στην πόλη μου θα πρέπει να μπορεί να ζεσταθεί. Εγώ δεν μπορώ να δεχτώ κάποιο να πεθάνει από το κρύο στην πόλη μου, είτε είναι κάτοικο τη πόλη μόνιμο, είτε είναι περαστικό από την πόλη. Αφού εγκατέστησα λοιπόν το 2008 αυτή τη θερμενόμενη σκηνή, πήρα επιστολή από το γαλλικό κράτος που μου λέγανε λίγο πολύ «Μα είσαστε τρελός, έτσι θα προσελκύσετε χιλιάδες και χιλιάδες και θα δημιουργηθούν διάφορα προβλήματα ασφάλειας, υπάρχουν λαθροδιακινητές μεταξύ αυτών και είναι δικιά σας ευθύνη γιατί είναι στη δικιά σας πόλη και να ξέρετε ότι το κράτος νύπτει τα σχήρας του». Οπότε ήδη άρχισε αυτός ο φόβος. Εγώ όμως την εγκατέστησα και μάλιστα εγκατέστησα και μια δεύτερη για να χωρίσω τις γυναίκες από τους άντρες και για μερικά χρόνια έτσι συνεχίσαμε. Οι γιατροί του κόσμου ήταν παρόντες και αυτοί φρόντιζαν, πρόσφεραν φροντίδα και δουλέψαμε με την οργάνωση αυτή, τους γιατρούς του κόσμου, για να καταστήσουμε και τουαλέτες, για να μπορούν να έχουν επίσης και ε, πόσιμο νερό. Και υπήρχαν εθελοντές από οργανώσεις που οργάνωναν ταξίδια λίγο πολύ για να μπορούν να πηγαίνουν στα ντους, στα μπάνια των ε, γηπέδων ή αλλού για να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να εξυπηρετούνται. Όμως στη Γαλλία αυτό θεωρείται ε, παράβαση διότι υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν καταδικαστεί άνθρωποι επειδή ακριβώς πρόσφεραν τέτοια βοήθεια ε, στον κόσμο. Οι οργανώσεις όμως και θελοντές το κάνανε και εμείς ανοίξαμε τα γεωναστήρια, τα γήπεδα για να μπορούν οι άνθρωποι να πηγαίνουν και να πλένονται. Το κάναμε αυτό λοιπόν από το 2008 μέχρι το 2015 όπου είχαμε 40-50 ανθρώπους. Το καλοκαίρι του 2015, όπως έγινε και στην υπόλοιπη Ευρώπη, μας έφτασαν και εμά μαζικά πρόσφυγες. 40-50 τον Ιούλιο, 190 στα τέλη του Αυγούστου. Οι οργανώσεις πάλι ήρθαν και μας είπαν προσοχή εμείς ναι, να δίνουμε φαγητό και ρούχα για 40-50 ανθρώπους αλλά για 190 δεν μπορούμε. Και συνέχιζαν να έρχονται άνθρωποι κάθε μέρα. Τότε λοιπόν επευθύνθηκα στο κράτος. Τι μπορεί να κάνει η γαλλική κυβέρνηση, ρώτησα για να μας βοηθήσει, για να υποδεχτούμε τους ανθρώπους αυτούς, ώστε να μην βρίσκονται όλοι στο ίδιο σημείο αλλά να ανοίξουμε και άλλους χώρους και να υπάρξει μια κατανομή της υποδοχής παντού στην Γαλλική επικράτεια. Ε, δεν πήρα απάντηση λοιπόν. Και ακόμα δεν έχω πάρει ικανοποιητική απάντηση, παρόλο που υπήρξε κάποια πρόοδος ε, την περίοδο αυτή 2015-2016. Με αντιπροσώπους από την Καρκουάς πήγαμε στον Υπουργό το Σεπτέμβριο του 2015 και ο Υπουργός είχαν μετρήσει και βρήκαν ότι δεν ήταν 190, ήταν 145. Δεν είχαν όμως ούτε οι τίποτα, ούτε να πληθούν, τουαλέτες. Έβρεξε και πολύ εκείνο το χειμώνα του 2015, δεν έκανε τόσο πολύ κρύο, αλλά έβρεξε πάρα πολύ. Και έτσι ο χώρος αυτός ήταν ένα έλος λασπόδες με 300 ανθρώπους, γυναίκες, παιδιά που παίζανε εκεί. Εγώ τρεπόμουν για αυτή την κατάσταση. Δεν μπορούσα να δεχτώ ότι είναι αυτός τρόπος υποδοχής των ανθρώπων. Πάλι ήρθα σε επαφή με τον Πρωθυπουργό τότε, με επιστολή μου, πρώτη, δεύτερη, τρίτη και ποτέ δεν πήρα απάντηση από τον Μανουέλ Βάλ στον Πρωθυπουργό τότε. Απευθύνθηκα, στο, στον ε, Πρόεδρο, πήρα μια τεχνοκρατική απάντηση που λίγο πολύ το ίδιο μου είπε, ότι δηλαδή δεν υπάρχει λύση. Από τους 145 τέλη Σεπτεμβρίου φτάσαμε 1200 τον Οκτώβριο, 2.500 το Δεκέμβριο. Χωρίς όμως να υπάρχει καμία βοήθεια, ούτε οικονομική ούτε τίποτα. Ήρθανε κάποια όργανα της τάξης κάποια στιγμή για να εμποδίσουν να έρχεται περισσότερος κόσμος, αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι αυτό είναι πολύ δύσκολο, άρα η καταστολή δεν είναι λύση, δεν βοηθάει. Είχαμε τα όργανα τη τάξη λοιπόν που ήρθαν και στις 13 Νοεμβρίου με αυτά που έγιναν στο Παρίσι, στο Πατακλάν κλπ. Τα όργανα τη τάξη πήγαν αλλού. Είχαν άλλη αποστολή και άρα μείναμε μόνοι μας. Και ο κόσμος συνέχιζε να φτάνει. Ακόμα και σήμερα, τον Ιούνιο του 2017, δεν υπήρξε καμία περίπτωση ε, Δηλαδή δεν συνέβη τίποτα, γιατί πολλά ακούμε για τους ανθρώπους αυτούς ότι υπάρχει ανασφάλεια, ότι είναι απαταιώνες λοιπά. Τίποτα. Δεν είχα κανένα τέτοιο περιστατικό όλα αυτά τα χρόνια. Τίποτα. Καμία τέτοια περίπτωση αδικήματος ε, στην πόλη. Το κράτος λοιπόν δεν έκανε τίποτα, δεν είχε και κανένα σχέδιο ούτε για να εμποδίσει την άφηξη, ούτε για να βοηθήσει τους ανθρώπους που ήδη βρισκόντουσαν εκεί. Οπότε ζήτησα από τους γιατρούς του κόσμου να σκεφτεί κάτι για το σχεδιασμό ενός καταβλισμού βάσει των αρχών του ΟΗΕ. Ξέρετε ότι όταν ε, συγκεντρώνονται πολλοί άνθρωποι μαζί πρέπει και δίπλα να υπάρχουν υποδομές για να πλένονται, να έχουν πόσιμο νερό, τουαλέτες κλπ. Είχαμε 2.500 λοιπόν όπως σας είπα το Δεκέμβριο και είχαμε προβλέψει σκηνές για 5 άτομα. Καταλαβαίνετε ότι ο Δήμαρχος δεν είναι σε θέση, δεν έχει τις γνώσεις να το κάνει αυτό σε χώρες που έχουν τη συνήθεια με ε, καταβλισμούς ίσως. Γι' αυτό και απευθύνθηκα λοιπόν στους ε, γιατρούς του κόσμου να οργανώσουν τέτοιες σκηνές για πέντε άτομα και γιατί για πέντε άτομα για να διατηρηθεί αυτός ο οικογενειακός πυρήνας. Οπότε 500 τέτοιες σκηνέ έπρεπε να δημιουργηθούν στην περιοχή για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να βολευτούν. Προβλέψαμε και μία συνέντευξη τύπου στις 23 Δεκεμβρίου του 2015. Στις 22 Δεκεμβρίου το βράδυ, στις 8, ο νομάρχης μου τηλεφωνάει και μου λέει μόλις με πήρε ο Υπουργός πριν φτιάξετε τον καταβλισμό αυτόν πρέπει να μιλήσετε μαζί του. Του είπα, μα δεν μπορώ να δω τον Υπουργό. Πριν αύριο έχω την συνέντευξη που μου είπε να πάτε στο Υπουργείο γρήγορα. Δέχτηκα λοιπόν, ανέβαλα τη συνέντευξη τύπου, πήγα για να δω τι έχει να μου πει ο Υπουργό. Οπότε, πολύ περιορισμένα με το σύμβουλό του, με ελάχιστου ανθρώπου δηλαδή. Του έδειξα τα σχέδια της πόλης και του είπα να, εδώ βρίσκονται 2.500 πρόσφυγες, να που θέλω να τους βάλω για να διασφαλίσω την αξιοπρέπειά τους. Γιατί πρόκειται για ανθρώπους, είτε είναι μετανάστες, είτε είναι πρόσφυγες, είτε όπως θέλετε ονομάστε τους, είναι άνθρωποι και θα πρέπει έτσι να τους συμπεριφερόμαστε. Και είναι αλήθεια ότι ο χώρος που είχα διαλέξει Εντάξει, ήταν ανάμεσα στις δρομικέ γραμμές και τον αυτοκινητόδρομο. Δεν ήταν τέλειο, αλλά ήταν η καλύτερη περίπτωση στην πόλη για να δημιουργηθεί ο καταβλισμό αυτό. Και είχαμε συνεργαστεί με οργανώσεις και είχαμε βρει λοιπόν ένα χώρο που δέχονταν και οι ίδιοι πρόσφυγες. Γιατί έπρεπε βέβαια θελοντικά να μεταφερθούν από το χώρο που βρίσκονταν στον καινούριο που θα φτιάχναμε. Οπότε έπρεπε να του κάνει και όσο φτιάχναμε τον καταβλισμό πηγαίναμε τους πρόσφυγες για να δούνε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τους ετοιμάζαμε να ζήσουν. Στη συνάντηση αυτή λοιπόν με τον Υπουργό Εσωτερικών εγώ πήγα με διάφορα επιχειρήματα νόμος για την υποδοχή παράνομων, το ήξερα ότι υπάρχει, αλλά βλέπετε στο Δήμο μου έχουμε και άλλους κώδικες που είναι δημοσίας υγείας, οικογένειας, που υποχρεώνουν τον Δήμαρχο να φροντίσει, να προσφέρει κάποια πράγματα σε αυτούς που βρίσκονται στην επικράτειά του, είτε πρόκειται για μόνιμους κάτοικους, είτε πρόκειται για περαστικούς. Οπότε, εγώ είπα, αν πρέπει να μου κάνουν δίκη, ωραία, να δούμε τελικά ποιο από του δύο κώδικε θα υπερισχύσει. Θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε ποια είναι η ιεράρχηση των ε, νόμων που ισχύουν. Οπότε, έτσι κι αλλιώς το κράτος και η πόλη του Καλέ έχει ήδη καταδικαστεί, γιατί δεν πρόσφεραν ε, τις υπηρεσίες που θα έπρεπε να μαζεύουν, τα σκουπίδια, να προσφέρουν ε, υποδομή για να πλένονται οι άνθρωποι να του υποδέχεται εξωπρεπώς. Και εγώ είπα ότι εγώ δεν θέλω το διοικητικό δικαστήριο να με καταδικάσει όπω έκανα με το καλέ επειδή δεν διέθεσα τι υποδομέ αυτέ στου ανθρώπου, και ούτε θέλω και τέτοιε συνθήκε ε, ζωή αναξιοπρεπή για του πρόσφυγες. Ο υπουργό ζήτησε από τον Μάρκ λοιπόν που με συνόδευε να δει με μένα ποια είναι τα προβλήματα που τίθενται. Γιατί πανέλα «Ναι, θα είναι πολύ κοντά στον αυτοκινητόδρομο, θα εμποδίζουν το αυτοκίνητο, θα είναι πολύ κοντά στι δρομικέ γραμμέ, θα μπλοκάρουν τα τρένα, την τοπική οικονομία, ε, οι πυροσβέστε, αν πρέπει να παρέμβουν, πώ θα κάνουν. Ήταν ένα χώρο κενό, έτσι. Λοιπόν, τέλο πάντων μου βάλανε ένα σωρό προβλήματα για να δυσκολέψουν την ε, δημιουργία αυτού του καταβλισμού, οπότε μου είπανε να ψάξω να βρω με τον ονομάρχη λύσεις όλα αυτά τα προβλήματα, τα οποία ο ονομάρχης όλο και έβαζε στο τραπέζι. Μέχρι τις 10 Ιανουαρίου δούλεψα λοιπόν με τους αστυνομικούς, τους πυροσβέστες, τις υπηρεσίες των συνδρομικών υπηρεσιών κλπ. κλπ. για να λυθούν όλα αυτά. Και 11 Ιανουαρίου πήρα γράμμα από τον Ομάρχη που είπε ότι δεν συμφωνούσε ακόμα με τη δημιουργία αυτού του ε, καταβλισμού γιατί θα προσέλκει και άλλους πρόσφυγες. Αλλά δεδομένων των απαντήσεων που εγώ του έδωσα σε όλα του τα επιχειρήματα, είπε ότι δεν θα με εμπόδιζε και να το κάνω. Δηλαδή, με λίγα λόγια έλεγε ότι δεν συμφωνώ μεν, αλλά άμα θέλετε να το κάνετε, κάντε το. Οπότε αρχίσαμε να οργανωνόμαστε, να φτιάξουμε αυτό τον καταβλισμό, φτιάξαμε ε, μια διαδρομή στη μέση, ε, να καθαρίσαμε, βάλαμε τουαλέτες, ντους, οι γιατροί του κόσμου επίσης βοήθησαν πολύ με σκηνές που εγκατέστησαν έβαλαν 120 σκηνέ. μετά είχαμε κατακλυσμό, έβρεξε πάρα πολύ και δυστυχώ καταστράφηκαν οι σκηνέ αυτές. Φτιάξαμε μετά κάτι ξύλινα σπιτάκια με πέντε θεσει Με 384 τέτοια σπιτάκια άνοιξε λοιπόν ο καταβλισμός εν τέλει. Ήταν μια παλιά αγρικία έτσι. Οπότε στο κτίσμα αυτό οργανώσαμε υπηρεσίες υγείας. Οι γιατροί του κόσμου, οι γιατροί χωρίς ε, σύνορα, οι γυναικολόγοι χωρίς σύνορα, οι γιατροί χωρίς σύνορα, όλοι αυτοί να μπορούν να βοηθούν τον κόσμο που έχει προβλήματα. Πήγανε 7 Μαρτίου οι πρώτοι κάτοικοι του καταβλισμού αυτού. 7, 8, 9 Μαρτίου σε τρει μέρες μετακόμισαν όλοι όσοι ήταν στον παλιό καταβλισμό πήγαν στον καινούριο. Τη στιγμή τη μετακόμισή, ο Νομάρχη εμποδίζει τα λεωφορεία που είχαμε στη διάθεσή μα να μεταφέρει τον κόσμο. Γιατί λέει τα λεωφορεία δεν ανταποκρίνονται στους ε, διάφορου κώδικε που ισχύουν για την ε, φωτιά και και τον κώδικα χωροταξία. Και γιατί το είπε αυτό, εμείς είχαμε σκηνές. Όταν έχουμε σκηνές δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ανταποκριθούμε στον κώδικα χωροταξία. Όμω, όταν υπάρχει κάτι πιο σταθερό, όπω ήταν αυτά τα ξύλινα σπιτάκια, τότε είπε Α, πρέπει να έχετε ε, ανοιχνευτή φωτιά. Ε, πρέπει να μπορεί τρία λεφτά να αντισταθεί το κάθε σπιτάκι στη φωτιά. Ε, Εμεί δεν τα είχαμε φροντίσει όλα αυτά, οπότε ήθελε να εμποδίσει τη μετακόμιση. Πήγα να δω τους ε, αστυνομικούς, οι οποίοι εμπόδιζαν την αναχώρηση των λεωφορείων και ρώτησα ποιο είναι το νομικό επιχείρημα που εμποδίζει τα λεωφορεία να φύγουν από τον παλιό καταβλισμό να πάνε στο καινούριο. Ο Νομάρχη είχε δυσκολευτεί γιατί δεν είχε επιχειρήματα, άφησε τα λεωφορεία λοιπόν να μετακινηθούν και έγινε μετακόμιση τι τρει αυτέ μέρε και πήγε καλά. Ήταν μια από τι πιο δυνατέ στιγμές τη ζωής μου να βλέπω τα παιδιά να πηγαίνουν πια στον καταβλισμό αυτό που μπορούσαν να παίξουν ποδόσφαιρο, να παίξουν ρακέτε, να ζουν τέλο πάντων κάτω από καλύτερε συνθήκε. Θέλαμε ο καταβλισμό αυτός επίσης να φυλάσσεται 24 ώρε στις 24 σε 7 μέρες τη βδομάδα. Και γιατί? Γιατί γνωρίζαμε ότι υπήρχαν λαθροδιακινητές. Δεν είναι οι καταβλισμοί που κάνουν τους διακινητές. Είναι η τύχη, τα σύρματα είναι η ελευθερία που προσελκύει τους πρόσφυγες και τους μετανάστες στις χώρες μας. Η Ευρώπη είναι η πρώτη οικονομία στον κόσμο. Στις χώρες τους δεν έχουν τίποτα. Δεν είναι οι καταβλισμοί που οργανώνουμε εμείς που προσελκύουν πρόσφυγες. Υπήρχε ένας με τον οποίο έπινα κάθε μέρα τσάι και μου είπε ότι μια μέρα είπε, μάλλον και μου είπε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόσφυγα ο οποίο λέει στη γυναίκα: Λοιπόν, σήμερα φτιάξα τη βαλίτσα σου, θα πάμε στην Grand Sand, εκεί θα μα υποδεχτούν καλά. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Το μόνο που υπάρχει είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να φύγουν από τι χώρε του που έχει πόλεμο, τρομοκρατία ή να φύγουν και από τι οικονομικέ δυσκολίε που αντιμετωπίζουν και που όταν κανεί έχει γυναίκε και παιδιά να θρέψει, θέλει να πάει να βρει δουλειά εκεί που υπάρχει δουλειά. Ισχύει αυτό παντού στον κόσμο. Οπότε εγώ δεν βάζω του ανθρώπου αυτού σε κατηγορίε. Η μετάβαση, σε πάση περιπτώσει, έγινε και αντί για 2.500 ανθρώπου είχαμε 1.300. 1.200 χάθηκαν ανάμεσα στο Δεκέμβριο και το Μάρτιο. Πήγαν στην Αγγλία. Μέσω Βελγίου ή Ολλανδίας που δεν είχαν προστατεύσει τα λιμάνια τους όπως το είχαμε κάνει εμείς στη Γαλλία και έτσι πολλά δίκτυα πήγαν από βελγικά και ολλανδικά λιμάνια. Οπότε όταν τελείωσε η μετακόμιση αυτή είχαμε 1.300 πρόσφυγες οι οποίοι καταστάθηκαν στο νέο μας καταβλισμό. Αρχίσαν εκεί τη νέα τους ζωή στην Grand Sand. Επαναλαμβάνω ότι εμείς στη Γαλλία και γενικά στην Ευρώπη δεν έχουμε εμπειρία με τέτοιους οργανωμένους καταβλισμούς Εμεί είπαμε στου γιατρού του κόσμου, δεν θέλουμε να είναι μια φυλακή, να μην υπάρχουν έλεγχοι στην είσοδο, να μην υπάρχουν ε, σειρματοπλέγματα γύρω-γύρω, να μην είναι σαν φυλακή. Και όντω αυτό κάναμε. Και έτσι λειτουργήσε. Και λειτουργήσε καλά. Μέχρι τον Αύγουστο. Υποδεχτήκαμε λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους, τους φροντίσαμε, ενώ στο παλιό καταβλισμό υπήρχαν προβλήματα με ασθένειες, πνευμονία οι άλλες οι οποίες είχαν εξαφανιστεί ουσιαστικά από τη Γαλλία αλλά εμφανίστηκαν και πάλι, τους λίγους μήνες που λειτουργήσε ο καταβλισμός αυτός, όλες αυτές οι ασθένειες εξαφανίστηκαν. Οι γιατροί του κόσμου, μάλλον οι γιατροί χωρί σύνορα, είπε κάποια στιγμή δεν έχουμε κανένα λόγο να βρισκόμαστε πια εδώ. Θα πάμε αλλού που υπάρχουν περισσότερε δυσκολίε είτε στη Γαλλία είτε αλλού στον κόσμο. Και μείνανε μόνο οι γιατροί του κόσμου. Τον Αύγουστο μας είχαν μείνει μόνο 700. Από τους 1.300 μείναμε στους 700, χωρίς ε, έλεγχο. Κάποιοι πήγαν στην Αγγλία, όπως συνεχίζουν ακόμα, και άλλοι που δεν θέλανε να υποβάλουν αίτηση ασύλου δεδομένων των συνθήκων που τους είχαμε υποδεχτεί με τη λάσπη, με αστυνομικού παντού χωρίς κανείς να νοιάζεται για αυτούς, κανένας δεν είχε ζητήσει άσυλο, με το νέο καταβλισμό 700 ζήτησαν άσυλο και έτσι μεταφέρθηκαν σε άλλους καταβλισμούς όπου βρίσκονται οι αιτούντες άσυλο. 700 λοιπόν μας μείναν τον Αύγουστο μέχρι τον Οκτώβριο, μέχρι που το γαλλικό κράτος αποφάσισε να διαλύσει αυτό που ονομάζαμε τη ζούγκλα του Καλέ. Μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο μέσα δεχτήκαμε άλλους 400 και το Δεκέμβριο αρχές Ιανουαρίου ήμασταν και πάλι 1500 στον καταβλισμό. Και πάλι δεν τους προσέλκυσε ο καταβλισμός ο δικός μας, είναι γιατί κλείσανε άλλες περιοχές, άλλοι χώροι όπου βρίσκονταν οι άνθρωποι αυτοί. το 2015-2016 σίγουρα υπήρξε πρόοδος. Όταν εγώ τον Αύγουστο αντιμετώπισα το πρόβλημα υπήρχε ένας καταβλισμός. Σήμερα είναι 500. 500 κέντρα υποδοχής σε ολόκληρη τη Γαλλία. Και αυτό που κάνω εδώ σήμερα εδώ σε εσά, το κάνω παντού όπου μου ζητούν να έρθω και να διηγηθώ τι έγινε στην Grand Sand και λέω ότι πολλοί δήμοι, πολλές ε, πόλεις στη Γαλλία δημιούργησαν ε, κάτι τέτοιο και όλοι οι δήμαρχοι μου λένε το ίδιο. Μου λένε μια χαρά τα πάνε με το, τους ντόπιου. Από όποιο πολιτικό κόμμα και αν είναι ο δήμαρχος, είτε από τη δεξιά είτε από την αριστερά, εντάξει δεν μιλάω για την άκρα δεξιά, όλοι μου είπανε, μα πάνε μια χαρά τα πράγματα. Το Σεπτέμβριο που μας πέρασε ήμουνα στην Χάβρη και εκεί μίλησα με τον σημερινό πρωθυπουργό και τότε με τον δήμαρχο και μου είπανε ότι μια χαρά πάνε τα πράγματα. Ελπίζω λοιπόν και η νέα κυβέρνηση να οργανώσει αντίστοιχα. Με 6.000 εθελοντές δουλέψαμε, πάνω από 50 οργανώσεις μη κυβερνητικές, Α, Κάτι είπα για τους λαθροδιακινητές. Θα επανέλθω γιατί είναι σημαντικό. Στο παλιό καταβλισμό, όταν άρχισαν να μας στάνουν πολύ μαζικά, φτιάξαμε κάποια μπάγκαλος με τουαλέτες και ντους το πρωί. Το βράδυ, όμως, κλει... βρισκόντουσαν κλειδωμένες ε, οι εγκαταστάσεις αυτές και αυτοί που τις φύλασαν ζητούσαν λεφτά από τους πρόσφυγες για να έχουν πρόσβαση. Πράγμα που σημαίνει ότι χρειάζεται να υπάρχει έλεγχος από τις αρχές ακριβώς για να αποφύγουμε τέτοια δίκτυα τα οποία αποτελούν μια γάγκρενα. Η... Μετά τα ναρκωτικά και τα όπλα, η τρίτη μεγαλύτερη λαθροδιακίνηση είναι ακριβώς αυτή των προσφύγων και των μεταναστών που έχουμε στον κόσμο. Μέχρι τον Απρίλιο του 2017, γιατί έπιασε φωτιά τον Απρίλιο, 33 δίκτυα τέτοιων λαθροδιακινητών συλλάβαμε. Και έτσι αυτό μας επέτρεψε να τους πιάσουμε και πολλές φορές καταδικάστηκαν με πολύ βαριές ποινές. Επίσης είχαμε πολλούς Κούρδους, είτε από τη Συρία, είτε από το Ιράν, είτε από το Ιράκ. Δεν είχαμε Αφρικανούς, από το κέρας της Αφρικής, ενώ υπήρχαν πολλοί τέτοιοι στο Καλέ, από το Σουδάν, την Ερυθρέα κτλ. Εμείς όχι, στην Grand Sand δεν είχαμε τέτοιους. Και ούτε είχαμε ανθρώπους από το Αφγανιστάν. Όλοι αυτοί μας ήρθαν από τον Νοέμβριο και το Δεκέμβριο που πήγανε στο Καλέ πρώτα και αυτό άρχισε να δημιουργεί εντάσεις. Δεν ήξερα ότι υπάρχουν κοινότητες που δυσκολεύονται να συνεπάρξουν. Η Κούρδοι και Αφγανοί. Έμαθα πολλά πράγματα από ανθρωπολόγους ε, αργότερα. Ε, χωρίζουν τις κοινότητες ακριβώς για να μην ε, υπάρχουν συγκρούσεις μεταξύ τους. Δουλέψαμε λοιπόν για μήνες, τα παιδιά πηγαίνανε σχολείο στα σχολιά της πόλης, άνοιξαν άλλα τρία και γυμνάσιο και λύκειο. Κάποιοι ανήλικοι έφτασαν στο Πανεπιστήμιο στη Δουκέρκη τώρα και συνεχίζουν τι σπουδέ τους. Όλα λοιπόν πήγαν πάρα πολύ καλά και όλα πήγαν πάρα πολύ καλά και με τους ντόπιου. Από την αρχή, από τον Αύγουστο, εγώ άρχισα να γράφω κάθε μήνα σε όλους τους κάτοικου της πόλης για να τους εξηγώ ποια είναι η κατάσταση, από πού μας ερχόντουσαν οι άνθρωποι αυτοί, τι διαδρομή είχαν ακολουθήσει, γιατί φεύγαν από τη χώρα του. και σιγά σιγά τους εξηγούσε όλα τα διαβήματα που έκανα στον Υπουργό, στον Πρωθυπουργό, στον Πρόεδρο, τι αρνητικές απαντήσεις έπαιρνα από όλους αυτούς και τι σχέδια είχαμε για τον καταβλισμό αυτό. Ένα μισή εκατομμύριο ξόδεψε η πόλη για να δημιουργηθεί αυτός ο καταβλισμός και 2,5 εκατομμύρια πήραμε από τους γιατρούς του κόσμου. Εννοείται ότι ποτέ δεν αποζημιωθήκαμε, αλλά για μας η αξιοπρέπεια των ανθρώπων αυτών μετρούσε περισσότερο. Το κράτος όμως που δεν ήθελε να ανακατευτεί καθόλου, 30 ε, Μαΐου ήρθαν για να υπογράψουν μια σύμβαση. Γιατί για να λειτουργεί 24 ώρες το 24 ώρο ένας καταβλισμός χρειάζεται πολύ κόσμο και δεν φτάνανε οι εθελοντές, δεν θα μπορούσαμε να βασιζόμαστε μόνο στους εθελοντές. Θα έπρεπε να υπάρχουν και μισθωτοί, οι οποίοι θα κάνουν την καθαριότητα, τη φύλαξη να υπάρχουν ε, και ε, υπηρεσίες ασφάλειας. 5 εκατομμύρια το χρόνο. Ήρθε λοιπόν το κράτος για να αναλάβει το κόστος αυτός. Κάτι που σημαίνει ότι άρρητα αναγνωρίζει το κράτος τη λειτουργία του καταβλισμού αυτού. Συνεχίσαμε λοιπόν από το Δεκέμβριο πέρυσι, δεδομένου ότι είχαμε όλο και νέους, και πάλι έγραψα στο κράτος ήταν κάπου 200-300 που θέλανε να φύγουν για κέντρα υποδοχή στην υπόλοιπη Γαλλία, αλλά το Παρίσι επίση είχε ανοίξει ένα καταβλισμό με κάπω διαφορετική λειτουργία. Πίεζε δηλαδή το κράτο. Έλεγε εμεί 5-10 μέρε του κρατάμε και μετά το κράτο θα πρέπει να του κατανείμει αλλού. Όλε οι θέσει που ελευθερώνονταν τελικά πιάνονταν από τον καταβλισμό αυτό του, του Παρισιού. Και έτσι εμεί δεν μπορέσαμε να κάνουμε τίποτα και αυξήθηκε ο αριθμός σε εμά μέχρι να αρχίσουν οι εντάσεις ανάμεσα στις κοινότητες μέσα στον καταβλισμό. Και τελικά κάηκε σε λίγες ώρες ολόκληρος ο καταβλισμός και αυτό οφείλεται σε ένα ξεκαθάρισμα ε, λογαριασμό μεταξύ Αφγανών και Κούρδων, λαθροδιακινητών και έτσι ό,τι είχαμε καταφέρει σε ένα χρόνο καταστράφηκε. Καταλαβαίνετε συναισθηματικά πόσο κόστησε αυτό σε όλους, στους εθελοντές, στους δασκάλους που είχαν υποδεχτεί στα σχολιά τους παιδιά, ε, στους ίδιους τους κατοίκους του καταβλισμού. Εγώ είδα έναν επιθεωρητή και συνεχάρη τους δασκάλους, τους καθηγητές, τους διευθυντές των σχολείων και όλοι κλαίγανε γιατί μας μετέφεραν τις εμπειρίες τους, την αλληλεγγύη που διαπίστωσαν μεταξύ των παιδιών, μεταξύ των γονιών και πόσο σημαντικό ήταν για τον Δήμο μας να ανοιχτεί στον κόσμο. Μερικές φορές είχα και παιδιά τεσσάρων ετών. Δημιουργήθηκε μια φοβερή οριμότητα για τα παιδιά αυτά που πιστεύω ότι τελικά βοήθησε. Ήταν μια καταπληκτική ανθρώπινη εμπειρία και νομίζω ότι όλοι όσοι πέρασαν από τον καταβλισμό όταν ε, έφυγαν από εκεί έφυγαν διαφορετικοί. Και πέρασαν πολλοί. Ε, και ευρωβουλευτέ, ξέρω ότι μας επισκέφτηκαν, βουλευτέ από τη Γαλλία, από τη Γερουσία, από τη Γαλλική Εθνοσυνέλευση, ε, τοπικοί εκλεγμένοι. Κάποιοι βουλευτές από την Πολωνία ήρθαν επίσης για να δούνε πώς λειτουργεί ο καταβλισμός αυτός, γιατί είχαν μάθει τα νέα στη χώρα τους. Ε, τα μέσα ενημέρωσης μας κάλυψαν πολύ. Και όλοι λοιπόν όταν βγήκαν από καταβλισμό ήταν διαφορετικοί. Και ο Υπουργό Εσωτερικών το είπε ότι ήταν άλλος άνθρωπος και Υπουργό ε, Κατοικίας όταν ήρθε για τη σύμβαση είδε ότι πρόκειται για ανθρώπινα όντα, ότι μπορούσαμε να μιλήσουμε μαζί τους, να ανταλλάξουμε απόψεις και ο Υπουργός πέρασε πολύ χρόνο μαζί τους. Στη βάση αυτή λοιπόν λέω ότι μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Σήμερα μας πετάνε νούμερα και μας λένε δεν μπορούμε να υποδεχτούμε εμείς όλη τη μιζέρια του κόσμου. 0,4% του ευρωπαϊκού ε, πληθυσμού είναι οι μετανάστες σήμερα. Τίποτα δηλαδή. Νομίζω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε και βλέπουμε ότι γίνεται. Αυτό που έγινε στη Γαλλία δείχνει ότι γίνεται. Και ζητάω από τη γαλλική κυβέρνηση να διευρύνει την προσπάθεια αυτή που έχει γίνει με τα κέντρα υποδοχής. Γιατί εγώ σήμερα αρχίζω πάλι να έχω 300 ε, ανθρώπους ε, πρόσφυγες ε, στην περιοχή μου, άρα αρχίζω την ιστορία πάλι από την αρχή. Γιατί δεν μπορώ να τους αφήσω έτσι. Πρέπει να τους προσφέρω αξιοπρεπείς συνθήκες. Φοβάμαι όμως ότι τώρα που πλησιάζει το καλοκαίρι θα μας αρχίσουν πάλι να έρχονται από την Αφρική και από αλλού και οι πρόσφυγες ξέρουμε και οι μετανάστες σήμερα ε, παίρνουν ακόμα μεγαλύτερο κίνδυνο για να έρθουν ε, στις χώρες μας. Διακινδυνεύουν πολύ περισσότερα, πληρώνουν πιο ακριβά το ταξίδι τους, γιατί είναι πιο δύσκολο. Εμείς πρέπει να συνεχίσουμε να τους υποδεχόμαστε. Η κρίση δεν είναι η κρίση του μεταναστευτικού, είναι της υποδοχής. Νομίζω ότι βρισκόμαστε στην αρχή και ότι θα έχουμε και άλλες εκατοντάδες χιλιάδες τα επόμενα χρόνια που θα μας έρθουν. Να λοιπόν ποια είναι η δικιά μου μαρτυρία που ήθελα να σας μεταφέρω σήμερα το πρωί και να σας πω ότι όταν εξηγούμε στον κόσμο, ο κόσμος καταλαβαίνει. Ξέρετε ότι έχουμε εκλογέ στη Γαλλία. Στον πρώτο γύρο Είμαι ο πρώτος δήμος ανάμεσα στη Δουκέρκη και την Λίλ, 80 χιλιόμετρα, που δεν έβαλε στο πρώτο γύρο των προεδρικών ε, εκλογών πρώτο κόμμα την άκρα δεξιά. Πολλοί κάτοικοι στην πόλη μου είναι περήφανοι για αυτά που κάναμε. Θέλησαν να συναντηθούν με τους ανθρώπους αυτούς, συναντήθηκαν και δεν μπορεί να είναι πολύ ευχαριστημένοι γιατί η οικονομία ενισχύθηκε. 46 θέσεις απασχόλησης δημιουργήθηκαν για αυτούς που έπρεπε να ασχοληθούν με τον καταβλισμό. Όταν δηλαδή η υποδοχή δεν γίνεται έτσι χαοδός αλλά οργανωμένα, μπορεί να λειτουργήσει πολύ καλά. Πιστεύω λοιπόν ότι μπορούμε να πολλαπλασιάσουμε τα κέντρα υποδοχής στη Γαλλία και εκ παραλίλου να δούμε πώς θα καταπολεμήσουμε τους λαθροδιακινητές, είτε με ανθρωπιστικές ε, διαδρόμους ε, άφηξης των ανθρώπων αυτών, είτε με θεωρήσεις, βίζα, που να μπορούν να πάρουν οι άνθρωποι αυτοί εκτός Ευρώπης για να έρθουν στην Ευρώπη. Εξάλλου, μπορεί να μην είναι ο πρώτος προορισμός των προσφύγων η Ευρώπη, είναι όμως ο πιο θανατηφόρος. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να κάνουμε κάτι για να μην συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Τελείωσα. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. <clears throat> Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ κύριε Καρέμ. Πολύ συγκινητικά αυτά που μας είπατε. Μπορώ να συνοψίσω. Ποιο είναι το πνεύμα των όσων μας είπατε. Πιστεύετε ότι οι άνθρωποι που είναι σε ηγετικές θέσεις θα πρέπει πραγματικά να ηγούνται. Αυτό είναι το μήνυμα. Um, but I... Αυτό θέλετε να πείτε. Ας ακούσουμε τώρα ερωτήσεις. Είμαι σίγουρος ότι έχετε. Ορίστε. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Ήταν πραγματικά ενδιαφέρουσα ερώτηση. Λυπάστε για κάποια πράγματα στον απολογισμό. Ε, λυπάστε για κάποια πράγματα. Έχετε μετανιώσει. Και ποιες συνέπειες του Brexit όσον αφορά την περιοχή σας, την πόλη σας. Είμαι Χριστίνα από τη Βαρκελόνη, δημοσιογράφος. Καμία λύπη δεν έχω, καμία, δεν μετανιώ για τίποτα θα μπορούσαμε να τα κάνουμε διαφορετικά, μπορούμε να μαθαίνουμε από αυτά που κάναμε. Αλλά ήταν τόσο όμορφη ε, περιπέτεια, περίπλοκη. Δεν κοιμήθηκα κι εγώ και οι υπηρεσίε μου, περάσαμε άϊπνε νύχτε, γιατί ήταν δύσκολα τα πράγματα, αλλά ήταν μια πολύ καλή περιπέτεια. Τι θα έκανε διαφορετικό. Το θέμα της συμπεριφοράς των κοινοτήτων και το μεταξύ των δύο φίλων ίσως η ελευθερία, η φιλελεύθερη συμπεριφορά θα ήταν κάτι που να αντιμετωπιστεί. Όπω είχαμε πρόβλημα του Κούρδου. Αυτό το λάμβανε υπόψη. Θα προστάτευα περισσότερο τι γυναίκε και τα παιδιά, του ευάλωτου, σε μία συγκατοίκηση. Κατά την άποψη των ΜΚΟ, γιατροί χωρί σύνορα, γιατροί του κόσμου κλπ ποτέ δεν είχαμε επιτόπου διαπιστωμένο βιασμό των γυναικών. Υπήρχαν διάφορα προβλήματα και βιοπραγίες στους δρόμους, αλλά όχι στα, στους καταβλισμούς. Υπήρχε φόβος. Είχαμε 1500 άτομα. Εγώ ήθελα να προστατεύσω την αξιοπρέπεια αυτών των ανθρώπων, αλλά έμαθα ότι συνέβησαν κάποια πράγματα που με αηδίασαν. Δεν τολμούσαν να πάνε στην τουαλέτα το βράδυ οι γυναίκες και φορούσαν επάνες γιατί φοβόταν να πάνε μόνο στην τουαλέτα το βράδυ θα το έκανα διαφορετικό για να τι προστατεύσω καλύτερα, για να μην έχουν κινδύνου που θα διατρέχουν. Κάποιε προσαρμογέ θα έκανα. Διαφορετικά δεν λείπουμε για κάτι. Το Brexit θα αλλάξει κάτι. Τι να πω τώρα. Δεν νομίζω. Κάτι μπορεί να αλλάξει βέβαια. Η προστασία της εργασίας στη Βρετανία οι Βρετανοί θέλουν να κλειστούν για να δώσουν στους Βρετανούς τις δουλειές τους. Αυτό θα σκληρύνει τους νόμους ε, πρόσβασης εργασίας στην ε, Βρετανία. Και αυτό δημιουργήσει και στους Ευρωπαίους πολλά προβλήματα. Ξέρω κάποιους Πολωνούς που εργάζονται αρκετοί από αυτούς στη Βρετανία και δεν ξέρω πώ θα κρατήσει και αν θα κρατήσει αυτό. Ε, για τους κοινοτικού ίσως να υπάρξει λύση, για τους άλλους είναι δύσκολα. Η σκλήρυνση τη πρόσβαση στην εργασία ίσω θέσει τροχοπέδι στη βούληση των ανθρώπων που θέλουν να πάνε στην Βρετανία. Ένα από του λόγου που θέλουν να πάνε στη Βρετανία αυτή ήταν ότι θέλαν να βρουν δουλειά. Δεν θέλανε να μείνουν αυτοί που μείνανε στο καλέ, να μείνουν στο καλέ, θέλαν να πάνε στη Βρετανία. Έπρεπε να τους αφήσουμε να σκεφτούν και όλα, να τους αφήσουμε κάποιο χρόνο να δούμε τι θα κάνουν να τους απαγορευτεί να πάνε στη Βρετανία. Είναι και το θέμα τη γλώσσα. Πολλοί μιλάνε αγγλικά και όχι τα γαλλικά. Άλλοι θέλουν δουλειά. Άλλοι θέλουν οικογενειακή επανένωση. Να βρουν εξαδέλφια, συγγενεί, γυναίκα, παιδί κλπ. Θείο, θεία που είναι στην Αγγλία. Αυτή είναι τις, οι λόγοι για τους να πάνε στη Βρετανία. Δεν ξέρω το Brexit θα δυσκολέψει τα πράγματα. Αν δυσκολέψει το να βρούνε δουλειά, θα επηρεαστούν και οι ροές που θα έχουμε εμείς και θα μένουν σε εμά. Αυτή τη συνέπεια βλέπω εγώ και φαντάζομαι που απορρέει από το Brexit. Το ίδιο συμφωνεί μεταξύ Βρετανίας ε, και Γαλλίας τα σύνορα τώρα στη Γαλλία, αν βάζαμε τα σύνορα στην Αγγλία δεν ξέρω τι θα γίνει. Από τη στιγμή που του βάζουμε στο καράβι και φτάνουν εκεί, του απαγορεύουν και του στέλνουν, πού θα του αφήσουν του ανθρώπου, στη μέση τη μάχη. Τι θα γίνει με την επιστροφή του. Υπάρχουν αλλαγέ μετά τη συμφωνία του Τουκέ. Δεν ξέρω τι θα γίνει, αν θα αλλάξει κάτι μέσω του Brexit. Έχω, θα έχουμε διαφορετικό τοπίο στο καλέ, δεν ξέρω. Αυτά είναι κάποιες, ε, αυτά είναι πρώτες σκέψεις που έχω. Ορίστε. Pierre Robert, Médecin du Monde, τους γιατρούς του κόσμου. Πώς έγινε η απαστικοποίηση της περιοχής. Πώς έγινε η επιλογή της στέγασης αυτών. Πώς έγινε η κατανομή αυτών των ανθρώπων στην περιοχή. Βέβαια είσαστε δήμαρχος. Δεν έχετε περιφερειακή αρμοδιότητα, αλλά τοπική της πόλης. Πώς βλέπετε την προσέγγιση που ακολουθήθηκε για την εγκατάσταση αυτών των ανθρώπων. Κοιτάξτε, το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε. Όταν παρήχθη το πρόβλημα, είχαμε 2.500 ανθρώπου. Όταν έκανε την επιλογή, δεν είχα 2.500 κατοικίε στην πόλη για να του το χάσω. Και γίνονται πιο περίπλοκα τα πράγματα για τι παρεμβάσει των ΜΚΟ και των διαφόρων φιλανθρωπικών οργανώσεων. Προβλήματα για την υγεία, για τη στέγαση, για τα τρόφιμα. Είπα ότι δεν είναι καλή λύση οι καταβλισμοί. Ήταν μια κατάσταση ε, κατεπίγουσα και πρέπει να αντιμετωπιστεί η ανθρωπιστική κατάσταση. Τι με καθησυχάζει και βλέπω πιο θετικά τα πράγματα. Πρώτα από το σύμφωνο του Άμστερνταμ που υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με αυτήν, η έννοια τη βιωσίμου πόλη πρέπει στα 14 θέματα να συμπεριλαμβάνει και την ενσωμάτωση, την υποδοχή των μεταναστών και των προσφύγων. Είναι καλό. Υπεγράφει στο Κίτο, στον Ισημερινό, ε, παρόμοια συμφωνία όσον αφορά τι μελλοντικέ πόλει για την υποδοχή μεταναστών και προσφύγων και νομίζω ότι είναι καλή λύση. Έχω ένα σχέδιο γειτονιά για στέγαση που θα ξεκινήσει αρχές του 2018. Σε αυτή τη στέγαση θα έχω ένα ποσοστό ε, κατοικιών για του μετανάστες. Κάνουμε και ανακαίνιση σε άλλη γειτονιά και θα έχω κάποιε κατοικίε που θα είναι υποδοχή μεταναστών και προσφύγων. Έτσι θα καταλήξουμε στι 36.000 κοινότητε στην ε, Γαλλία. Μια περιοχή σε κάθε κοινότητα θα αφιερώνεται σε αυτό. Μπορεί να έχουν περισσότερες τέτοιες γειτονιές σε μεγαλύτερες πόλεις. Θα δούμε πώς θα δημορφωθεί η κατάσταση και πώς θα λειτουργήσει αυτή η λύση. Γι' αυτό κάναμε καταβλισμό παρά υποδοχή σε κανονική μόνιμη στέγαση. Για λόγους ανθρωπιστικούς δεν είναι καλή λύση αυτή. Είναι πολύ καλύτερη άλλη η λύση που τους δίνουμε κάποια στέγαση σε κάποιες γειτονιές από ότι ο Σε καπόλος, από το Irish Times, ε, Δουβλίνο. Δύο ερωτήσεις. Πρώτη, περισσότερα μας λέτε στο τι έγινε στους πρόσφυγες μετά την πυρκαγιά. Πού πήγαν, πώς ρυθμίστηκε. Δεύτερον, αναφερθήκατε στις γυναίκες και πόσο ευάλωτες ήταν στους καταβλισμούς και που δεν ήθελαν να πάνε το βράδυ στην τουαλέτα. Ξέρω ότι αυτό έχει προκύψει σε πολλού καταβλισμού στην Ελλάδα και την Ιταλία. Μπορείτε να μα πείτε περισσότερα πράγματα, τι προσπάθειε πρέπει να γίνουν, ούτω ώστε οι γυναίκε αισθάνονται ασφαλέστερε στου καταβλισμού. Απάντηση. Όταν έγινε η πυρκαγιά, ανοίξαμε τι αθλητικά κέντρα στο κέντρο και δύο στι γειτονικέ πόλει και στεγάσαμε όλου που ήθελαν να πάνε. Το βράδυ της πυρκαγιάς από 1500 άτομα του καταβλισμού στεγάσαμε 800 με 900. Αυτούς που ήθελαν. Και τις επόμενες μέρες στεγάσαμε 1300 συνολικά. Τους τοποθετήσαμε όλους σε κέντρα υποδοχής στη Γαλλία. Ω διαθαύματο απελευθερώθηκαν 1.300 θέσει στη Γαλλία σε τέσσερι μέρε. Διοργανώσαμε λοιπόν την αναχώρηση με λεωφορεία σε όλη τη Γαλλία. Πήγαν αυτά τα άτομα, οικογένειε, και οι μοναχικοί άνθρωποι. Για κάποιου δεν υπήρξαν δυσκολίε, το δέχτηκαν αμέσω, για άλλου πρέπει να του πείσουμε. Διότι όταν διασχίσαν χιλιάδε χιλιόμετρα υπό δυσχερέστατε συνθήκε και φτάνουν στα 30 χιλιόμετρα από τη Βρετανία και δεν έχουν μπροστά του μόνο τη θάλασσα και του λέμε θα πάτε στη Λιόν, στη Μασαλία, στην Τουλούζη κλπ. Αυτό του απομάκρυνε το στόχο. Αλλά του λέγαμε δεν μπορείτε να μείνετε έτσι εδώ. Το δέχτηκαν να φύγουν και τους στεγάσαμε. 1.254 στεγάσαμε σε κέντρο υποδοχής. Και συλλάβαμε και 40 διακινητές. Όταν πήγαμε, με... πήγαμε στο κέντρο λοιπόν και τους είπαμε δεν μπορεί να μείνετε εσείς εδώ γιατί κάθε φορά που κάποιος δεχόταν να πάει σε κέντρο υποδοχής 10 με 12 χιλιάδες ευρώ ξέφευγαν από τους διακίνητες κάνανε, μας υπονομεύανε από πίσω αυτοί οι άνθρωποι που του εντοπίσαμε τελικά. Και μπήκαν αστυνομικοί με πολιτικά και τους ε, απομακρύνανε. Φύγανε, κάποιοι γύρισαν. Από τους 1200 που έφυγαν, καμία εκατοστή επέστρεψαν, όχι περισσότεροι. Όπως και στο Καλέ λίγο πολύ, από τους 4.000, 600 επέστρεψαν, όχι περισσότεροι από αυτούς. Αυτό σημαίνει ότι η τελική λύση ε, το κέντρο υποδοχή λειτουργήσε και τα δίκτυα διοργανώθηκαν διαφορετικά. Ήμουν σε επαφή με αρκετού από αυτού όσον αφορά τα κοινωνικά δίκτυα και κάποιοι που ήταν στι Άτε, στη Ρεν και αλλού. Ε, μετά από τρει μέρε μου είπαν ότι ήταν στη Βρετανία. Μετά τη ΣΑΤ οι Περέν διοργανώθηκαν για να πάνε προ την Βρετανία. Οπότε γίνεται σχεδόν ψευτοπρόβλημα ε, διότι ε, πιο μακριά γίνεται οργανώνονται τα περάσματα προ τη Βρετανία Πώς καταλαπολεμούμε το θέμα, το πρόβλημα των παιδιών και των γυναικών. Ίσως να έχουμε ειδικού τόπους για αυτούς. Αλλά ήταν ένα θέμα που θέσαμε και ΜΚΟ στην είσοδο του, του καταβλισμού. Όταν είχαν πολύ κόσμο και δεν μπορούσαμε να τους χειριστούμε σωστά, του είπα: Δεν παίρνουμε κανέναν άλλον. εκτός από γυναίκες και παιδιά, οικογένειες, Διότι είναι πιο ευάλωτοι. Αλλά οι ΜΚΟ μου είπαν ότι οι άντρε μόνοι του ε, είναι και αυτοί ευάλωτοι. Είναι δύσκολο να βλέπουμε ποια, ποιο είναι το επίπεδο του ευαλώτου χαρακτήρα του καθενός. Θα πρέπει να ασφαλίζουμε τους τόπους, τις διάφορες περιοχές, τους καταβλισμούς, θα πρέπει να υπάρχουν ειδικοί χώροι. Αυτό γίνεται σε καταβλισμούς που δεν ξέρω εγώ, αλλά ο Μισελ Αζιέ, ε, ένας άλλος Γάλλος εκπρόσωπος που έχει δει πολλά τέτοια, μου εξήγησε πώς γίνεται. Τι είδα αλλού. Όταν υπάρχει ένας καταβλισμός να έχουν ασφαλείς χώρους για τους ευάλωτους ανθρώπους αν έχουμε τώρα τις διάφορες κατοικίες και τις μικρότερες υποδομές θα δημιουργηθεί ε, ε, θα υπάρχουν πάλι προβλήματα αλλά δεν θα είναι τόσο διάχυτο όσο είναι στον καταβλισμό Άλλες ερωτήσεις Ελεονόρα Καμίλη Αγάσμο κοινωνικό φορέα ποια είναι η απάντηση του τόπιου πληθυσμού για τη δουλειά που έγινε υπέρ των προσφύγων διότι περιχύνει περιοχή καλέ αισθάνθηκε έντονα την επιρροή του Front National ε, και όλους τους λόγους, τους μισαλόδοξους που ακούστηκαν κατά των μεταναστών. Ποια ήταν η επιρροή στη δική σας περιοχή. Απάντηση. Ο πληθυσμός Αύγουστο-Σεπτέμβριο. Γίνανε γρήγορα τα πράγματα. Δεν τόλμησαν να πάνε στα... στους παλιούς καταβλισμούς. Για πολλούς από αυτούς πρέπει να πω ότι ανακάλυψαν αυτά που συνέβησαν στα στρατόπεδα από την τηλεόραση, οι κάτοικοι. Και είχα διάφορε αντιδράσει στο Δημαρχείο. Μου έλεγαν δεν μπορούμε να του αφήσουμε έτσι. Δεν μπορούμε να του αφήσουμε να ζουν εκεί που δεν θα βάλαμε καν τα σκυλιά μας να παίξουν. Άρα υπήρχε μεγάλη συμπάθεια, κατανόηση ε, για αυτού από πλευρά πληθυσμού. Λοιπόν, ανακοινώσαμε και τα μέτρα για την υποδοχή που θέλαμε να κάνουμε. Αυτό επηρέασε πολύ τον πληθυσμό. Ποτέ δεν είχα διαμαρτυρίε, ποτέ δεν είχα κάποια διαδήλωση ε, του πληθυσμού να μου πει πληθυσμό, διώξτε του, δεν αντέχουμε, απομακρύνετε του, συνοδεύστε του, στείλτε του στη χώρα του. Τι θέσει λοιπόν του εθνικού μετόπου, οι θέσει του εθνικού μετόπου δεν πέρασαν στον πληθυσμό. Ε, αυτά από αυτού που ήρθαν να με δουν. Ε, υπάρχει και σιωπηλή πλειοψηφία που δεν ξέρουμε τι σκέφτονται. Οι εκλογέ που έγιναν, οι προεδρικέ και ο πρώτο γύρο μου έδειξαν ότι τελικά η πλειοψηφία του πληθυσμού δεν ήταν κατά αυτό που κάναμε στι προσφυγέ. Είμαστε μόνη πόλη που είχε επικεφαλή στην αριστερή, ε, αριστερά στο, στον πρώτο γύρο. Αλλού ήταν το εθνικό μέτωπο που ήταν επικεφαλής. Άρα αυτό είναι ένα καλό μάθημα που μπορούμε να δείξουμε στους ε, δημάρχους που συχνά φοβούνται να κινηθούν σε αυτό το τομέα. Λοιπόν, η απάντηση θα δοθεί από του Δημάρχου. Πιστεύω ότι οι χώρε θα έχουν δυσκολίε να βρουν ένα πρόβλημα. Αληθεύει για την υποδοχή των προσφύγων, όπω την αλλαγή του κλίματο, ε, όπω και για πολλά άλλα πράγματα και άλλα προβλήματα στη Γαλλία, όπως σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες ισχύει αυτό, αλλά ισχύει και για το Δήμαρχο της Βαρκελόνης. Υπάρχουν πόλεις που πολεμούν κατά της αλλαγής του κλίματος, όπως ανέσυρε ο Τρόμπο θα αποσύρει τη ΣΥΠΑ, αλλά είπαν οι Δήμαρχοι Αμερικανικών πόλων, εμείς θα συνεχίσουμε. Οι λύσεις πιστεύω θα έρθουν από την τοπική αυτοδιοίκηση που θα κάνουν τα πάντα να εφαρμόσουν λύσεις και θα υποχρεώσουν τους ηγέτες τους, τους τις κυβερνήσεις να τεθήσουν αυτές τις λύσεις. Παρά τη θέλησή του ενδεχομένω. Έτσι θα λειτουργήσει πιστεύω το πρόβλημα. Εμένα μου αρέσει ένα βιβλίο που, έλεγε, που λέει αν οι δήμαρχοι κυβερνούσαν τον κόσμο. Η κυβέρνηση των δημάρχων. Ε, πρέπει να το έχουμε αυτό σαν έννοια υπόψη μας. Έχουμε τη δυνατότητα να τα κάνουμε αυτά, έχουμε άμεση επαφή με τον πληθυσμό και μπορούμε να εξηγήσουμε στον κόσμο ακριβώς τι συμβαίνει. Υπάρχει μια σχέση εμπιστοσύνης που υπάρχει ανάμεσα στο Δήμαρχο και στο Δήμο, στον πληθυσμό του Δήμου και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτή την εμπιστοσύνη για να προωθήσουμε αυτές τις ιδέες. Άλλες ερωτήσει. Ορίστε. Έχω μια τελευταία ερώτηση. Εγώ, αν δεν έχει υπάρχει άλλος. Α, εσείς, ορίστε. Ποια είναι η κατάσταση σήμερα στο Grand Saint. Έχουμε και πάλι πολλούς μετανάστες που έρχονται, αλλάζουν τα πράγματα καθημερινά. Υπάρχουν μετανάστες που έρχονται στη Γαλλία μέσω Ιταλίας. Υπάρχει, έχουμε τη δευτεροβάθμια ε, μετακίνηση, δηλαδή επιστροφή μεταναστών από Γερμανία από αλλού. Απάντηση. Χθε είχαν περίπου 300 στην πόλη. Σε μια δασική περιοχή που έχουμε, μεταξύ του παλαιού και του νέου καταβλισμού, κάποιοι είναι άνθρωποι που ήταν στον καταβλισμό που ήρθαν ξανά, αλλά δεν είναι περισσότεροι. Για τους άλλους είναι περίπλοκο να που ήρθαν. Δεν έχουμε πλέον προσωπικό που να είναι παρόν μετά την πυρκαγιά του καταβλισμού ε, ε, δέχτηκα μεγάλο πλήγμα. Δεν ξανάρχισα από την αρχή γιατί είχαμε προεκλογική περίοδο. Ε, έπρεπε να σχηματιστεί η νέα κυβέρνηση για να έρθω σε επαφή με την κυβέρνηση για να δούμε ποια θα είναι η πολιτική για τη μετανάστευση. Από τη στιγμή που ο Υπουργό Εσωτερικών διορίστηκε, Τετάρτη στι 3 ώρα, 5, ξέρω εγώ πήρα τηλέφωνο στο Υπουργείο για να κλείσω ραντεβού. Μετά από 10 μέρε με κάλεσε για να μιλήσουμε τηλεφωνικά και όχι να μου δώσει ραντεβού. Το αρνήθηκα στην αρχή. Μετά συζήτησα με τον Ομάρχη λίγο αργότερα και τελικά δέχτηκα να ξανατηλεφωνήσω στον Υπουργό και την περασμένη Παρασκευή του μίλησα στο τηλέφωνο. Για την ώρα δεν μου μίλησε για, κατασπαρά, για καταστολή. Ε, για παρέμβαση τη Ευρωπαϊκή Ένωση για διαπραγμάτευση με τη Λιβύη για να κάνει ό,τι περίπου κάνει η Τουρκία να κάνει η Λιβύη. Δεν είναι αυτό λύση. Ε, μου είπε ότι θα αποστείλει δυνάμει τη τάξη, αλλά αυτό δεν είναι ούτε αυτό μου μίλησε μόνο η καταστολή και όταν το είπα κάθε φορά ότι αυτό δεν είναι λύση, βλέπετε πολύ καλά στην ιστορία τι συνέβη, σε μένα, στο Παρίσι και αλλού, αυτό δεν λειτουργεί, θα πρέπει να, αν υπάρχει καταστολή, τι κάνουν αυτού του ανθρώπου. Αυτό που συμβαίνει σήμερα στο Καλέ και αυτό που συμβαίνει σε μένα τι είναι, ότι έρχεται η αστυνομία, παίρνουν τις σκηνέ κλπ. Αλλά δεν παίρνουν τους πρόσφυγες, δεν τους συλλαμβάνουν, δεν έχουν τα μέσα να συλλάβουν 300 ανθρώπους και να τους οδηγήσουν δεν ξέρω πού διότι δεν μπορούν να το κάνουν. Δεν έχουν τα μέσα να το κάνουν, διότι ο νόμος δεν το επιτρέπει. Και εν πάση περιπτώσει δεν αποτελεί λύση. Λοιπόν, τους διασκορπίζουμε και ξανάρχονται. Και αυτό γίνεται επί εβδομάδε. Και νομίζω ότι θα διαρκέσει αν δεν υπάρξει πραγματική πολιτική που θα εφαρμοστεί και κυρίω όσον αφορά αυτό το κομμάτι τη Γαλλία γύρω από το καλέ. Διότι όσο η Βρετανία δεν θα μεταφερθεί στα ανοιχτά, θα έχουμε πάντα αυτό το πρόβλημα. Θα πρέπει λοιπόν και αυτό προτείνω στον Υπουργό. Θα πρέπει στον Κανσέντ να υπάρχει μια δομή με 100, να έχουμε 100 ανθρώπου στο καλέ, να υπάρχουν κάποιοι άλλοι 100 στην πουλών σειρμέων, να υπάρχει αλλού και αλλού να υπάρχει αλλού, εδώ, εκεί, αλλού, να κατανεμηθούμε γύρω από το καλέ, να υπάρξουν δομέ, να μπορούμε να έχουμε υποδοχή των ανθρώπων για κάποιε μέρε και μετά μετακινούνται. Όσο είναι εκεί δεν είναι αλλού όμω. Ε, λοιπόν, είμαστε χώρα κράτου δικαίου και πρέπει να εφαρμόσουμε τα δικαιώματα των ανθρώπων, να τα προστατεύσουμε και να σεβαστούμε την αξιοπρέπεια αυτών των ανδρών και των γυναικών που περνούν από την περιοχή μας. Ελπίζω ότι ο υπουργό ε, θα συνοηθεί. Δεν... Μόνο που μιλήσα στο τηλέφωνο κατάλαβα ότι δεν συμφωνώ αυτά μου προτείνει και πρότεινε κάποιο ραντεβού. Εγώ δεν θα περίμενα για πολύ. Δεν ανέχομαι αυτή την κατάσταση. η κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί, να έχουμε πολλού περισσότερου που θα καταφτάσουν. Δεν θέλω να ξαναζήσω το καλοκαίρι του 2015 στον Κανσέν. Θα πρέπει λοιπόν το γαλλικό κράτο να βιαστεί να εφαρμόσει κάποιε λύσει. Η κυβέρνηση δεν είναι πολύ ζεστή γι' αυτό, για το θέμα τη υποδοχή. Αλλά ο Πρωθυπουργό ήταν ευαίσθητο. διότι έχει την εμπειρία τη Χάβρη, ο Νίκολα Ιλό, ε, και αυτό είχε μπει στην κυβέρνηση, που έκανε κάποια παρέμβαση προ την κυβέρνηση, παλιά, ήρθε να επισκεφθεί τον Κανσέντ. Ήξερε γιατί πράγμα μιλάμε. Ίσως θα επηρεάσει ο Νικόλα Ιλουέ την κυβέρνηση για να διοργανωθούν κάπω τα πράγματα και να γίνει κάτι γρήγορα, γιατί πρέπει να κινηθούν πάρα πολύ γρήγορα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τα ειλικρινή σας λόγια, τη μαρτυρία σας. Νομίζω πως πραγματικά ήταν πολύ ενδιαφέροντα όσα ακούσαμε. Μας άνοιξαν τα μάτια για το πώς λειτουργεί η πολιτική. Τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ευρωπαϊκή νομοθεσία, όσο και σε τοπικό επίπεδο, που είναι πιο αληθινό, πιο πρακτικό. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Σας εύχομαι καλή συνέχεια Καλή δουλειά. I, uh, now... Λοιπόν, προτείνω να συνεχίσουμε με το επόμενο πάνελ. το οποίο θα συνεχίσει μέχρι τις 11 και 4. Εδώ έχουμε τους προσκεκλημένους από όλη την Ευρώπη, εσάς. Σας καλώ λοιπόν να έρθετε εδώ, να καθίσετε κοντά μου. Αυτό το πάνελ έχει ως θέμα τις προκλήσεις της ένταξης, εμπειρίες και ιστορίες από όλη την Ευρώπη. Αποφασίσαμε να κάνουμε ένα τέτοιο θέμα συζήτησης έτσι ώστε να μάθετε διάφορες εμπειρίες, να ακούσετε διάφορες ιστορίες από όλη την Ευρώπη. Όχι μόνο από τον Νότο, αλλά και από άλλα σημεία της Επίρου.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 Okay. I, uh, I invite you to take your seat. Παρακαλώ, καθίστε συνάδελφοι. Okay. Um, we, we, um, I, I'm, I'm a bit of a stickler on time. Λοιπόν, θα ήθελα να κρατήσουμε το χρονοδιάγραμμα, γι' αυτό λοιπόν προτείνω να αρχίσουμε. Να αρχίσουμε και διότι έχουμε φορτωμένο πρόγραμμα. Στις 11 και 4 περιμένουμε τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου και θα πάρει τότε το λόγο. Μετά αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε αν χρειαστεί τη συζήτησή μας. Αν θέλετε να κάνετε κάποιες ερωτήσεις παραπάνω, μπορείτε και μεταξύ σας να συνομιλήσετε. Μετά τις 12 όμως ε, δεν θα έχουμε τη δυνατότητα διερμηνίας, γι' αυτό λοιπόν πρέπει να εκμεταλλευτούμε το χρόνο που έχουμε. Αρχίζω λοιπόν με κάποια εισαγωγικά σχόλια. Στα αριστερά μου Έχουμε την Βιόλα Βίντερστάιν, συντονίστρια για θέματα ε, βοήθειας και ένταξης των προσφύγων από το Περιφερειακό Γραφείο του Βερολίνου των ε, Ιωαννητών. Μετά, ε, Πιέρ Βερμπέρεν, Γενικός Διευθυντής από τους Γιατρούς του Κόσμου Βελγίου. Στα δεξιά μου τον, ε, έχουμε τον Άντρα Κόβατς, διευθυντή του, της Οργάνωσης Προστασίας Προσφύγων Μέντεκ και την ε, κυρία Αγνές Ελάτσε, ερευνήτρια για ανάλυση πολιτικής στους τομείς της μετανάστευσης και ένταξης από το κέντρο προβίντου στη Ρήγα της Λετωνίας. Και επίσης ο κύριος Σταύρος Μυρογιάννης, διευθυντής και υπεύθυνο του ε, Καράτεπέ, στη Μητυλίνη, στη Λέσβο. Σκοπός αυτού του πάνελ είναι να μας δώσει τις διάφορες εμπειρίες ε, στην Ευρώπη. Ως συνέχεια των όσων μας είπε ο κύριος Καρέμ θα ακούσουμε τις μαρτυρίες για αυτά που γίνονται στο πεδίο και για το πώς εφαρμόζεται η πολιτική στην πράξη. Πώς περνάμε από τη θεωρία λοιπόν στην πράξη. Προτείνω λοιπόν να προχωρήσουμε ως εξής. Να ζητήσω καταρχάς από τους προσκεκλημένους να μας παρουσιάσουν ποιοι είναι, τι ε, κάνουν να παρουσιάσουν τις δικές τους μαρτυρίες και μετά θα έχετε το χρόνο να κάνετε τις ερωτήσεις σας. Μπορείτε λοιπόν τώρα να φορέσετε τα ακουστικά σας, διότι θα ακούσουμε διάφορες γλώσσες. Και θα ζητήσω λοιπόν από τους ομιλητές να είναι περιεκτικοί και σύντομοι. Καθώς και να μας μιλήσουν με κάθε ειλικρίνεια. Αρχίζουμε λοιπόν με τον κύριο Μυρογιάννη, αν συμφωνείτε. Έχετε το λόγο. Λέγομαι Σταύρος Μυρογιάννης και είμαι έρχομαι από την υπέροχη Λέσβο, από ένα ελληνικό νησί, από ένα ελληνικό νησί γεμάτο φιλοξενία και αλληλεγγύη. Σας μεταβιβάζω και φέρνω τους χαιρετισμού του Δημάρχου μας, του κ. Σπύρου Γαλινού, του προτεργάτη της φιλοξενίας μπορώ να πω γιατί για μας ε, η υπόθεση προσφυγικό και μεταναστευτικό είναι μια μεγάλη ευθύνη και μια μεγάλη υπόθεση φιλοξενίας. Αν πάρουμε το ρομαντικό κομμάτι του θέματος, ε, εγώ προσωπικά δεν είμαι καθόλου ρομαντικός, είμαι ρεαλιστής και βλέπω τα πράγματα face to face, στα μάτια που λέμε και εμείς οι Έλληνες. Αν πάρουμε λοιπόν το ρομαντικό, τη ρομαντική πλευρά του θέματος, νιώθουμε σαν πρεσβευτές και σαν αντιπρόσωποι της ευρωπαϊκής φιλοξενίας. Στο, στο καλωσόρισμά μου σε όλους τους α, επισκέπτες, τους λέω καλώς ήρθατε στην Ελλάδα, καλώς ήρθατε σε αυτό το υπέροχο νησί τη Λέσβο, με τις, το, τόσες, τις τόσες ομορφιές και τους υπέροχους κατοίκους, γεμάτους φιλοξενία και αλληλεγγύη, καλώς ήρθατε στην Ευρώπη. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί πολλά που είπε ο Δήμαρχος προηγουμένως ε, μπορώ να πω ότι τα αντιμετωπίσαμε και εμείς στο νησί μας. Τα αντιμετωπίσαμε και εμείς στην Ελλάδα, τα αντιμετωπίσαμε, τα αντιμετωπίσαμε και εμείς σε ένα ευρωπαϊκό έδαφος. Όταν λοιπόν λέμε ότι δίνουμε την πρώτη φιλοξενία των Ευρωπαίων πολιτών, νιώθουμε μεγάλη ευθύνη για αυτό που σηκώνουμε στις πλάτες μας. Ε, τα προβλήματα μεγάλα και σοβαρά δεν είχαμε μεγάλες διαφορές με το Καλέ και με τις άλλες πόλεις. Ευτυχώς εμείς ε, μπορέσαμε και πήραμε τα πράγματα στα χέρια μας πολύ γρήγορα από τον ε, Απρίλιο του 2015 που άρχισε η κρίση, η υπόθεση φιλοξενίας σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που είχαν ε, ανάγκη να φιλοξενηθούν ζητώντας άσυλο και άλλες υποθέσεις, υποθέσεις επανασύνδεσης με τις οικογένειές τους από τον Απρίλιο του 2015, αυτό μέχρι τον Οκτώβριο του 2015, ζούσαμε σε μια κόλαση. Όσο παράξενο και να σας φαίνεται. Κανένας δεν είχε προβλέψει, αν και γνωρίζαμε, γνωρίζαμε όλοι, γενικά, όχι εμείς που ζούσαμε στη Λέσβο, και δυστυχώς δεν είχαμε πάρει τα απαραίτητα μέτρα για να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση τέτοια μεγάλης άφηξης επισκεπτών, ταξιδιωτών που αυτοί οι άνθρωποι θα είχαν μεγάλε ανάγκε, ανάγκε υγεία, ανάγκε βιοπορισμού, ανάγκε καθημερινότητα. Αυτά που προανέφερε προηγουμένω ο κύριος Δήμαρχος, ε, βρίσκω σε αυτά που προανέφερε, βρίσκω πάρα πολλέ ομοιότητε με το δικό μα νησί, με τη δική μα υπόθεση. όμω όμως από 4-5 μήνε αλλάξαμε σχεδόν τα πάντα με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βεβαίως, με την ε, αρρωγή και τη βοήθεια των μη κυβερνητικών οργανώσεων και οργανώσεων και λίγο μπορώ να πω, ναι βεβαίως, μάλλον και τη βοήθεια του επίσημου ελληνικού κράτους. Γυρίσαμε τα πράγματα, γυρίσαμε την κόλαση στην αξιοπρέπεια, στην κανονικότητα. Σχεδιάσαμε ένα καινούριο κέντρο και βασίσαμε όλο το πλάνο και τη στρατηγική πάνω σε τέσσερις λέξεις. Αυτές οι λέξεις είναι ελευθερία, δημοκρατία, σεβασμός, αξιοπρέπεια. Πάνω λοιπόν σε αυτές τις τέσσερις λέξεις χτίσαμε αυτό το οικοδόμημα που λέγεται Καράτεπε. Μαυροβούνι. Κέντρο φιλοξενίας του Δήμου Λέσβου. Μια υπόθεση τοπικής εμβέλειας. Μια υπόθεση των τόπιων. Μια υπόθεση των κατοίκων, των δημοτών. Γιατί όπως σας είπα και πιο μπροστά, η φιλοξενία και η αλληλεγγύη είναι στο DNA μας. Δεν το ζορίζουμε καθόλου. Μας βγαίνει. Αγαπάμε τους, τον συνάνθρωπο. Αγαπάμε τους επισκέπτες. Θέλουμε να προσφέρουμε πολλά σε αυτούς. Δυστυχώς, στεναχωριόμαστε και θυμώνουμε όταν δεν μπορούμε να το κάνουμε. Ή αν υπάρχουν άλλοι παράγοντες που δεν μας αφήνουν να το κάνουμε. Παράγοντες πολιτικής δόξας, παράγοντες, οικονομικ... Ε, παράγοντες οικονομικοί, παράγοντες γενικά δόξας και διαφόρων παιχνιδιών πάνω στις πλάτες αυτών των ανθρώπων και στις δικές μας πλάτες. Εκεί μπορώ να πω να είμαστε αγνοί. Δεν, είχαμε, ε, δεν ήμασταν τόσο πονηροί ή μάλλον δεν γνωρίζαμε. Μετά όμως από δύο χρόνια μάθαμε. Ξέρουμε. Ξέρουμε να φιλοξενούμε πλέον αυτούς τους ανθρώπους που λέγονται πρόσφυγες και μετανάστες που για μας είναι φιλοξενούμενοι ταξιδιώτες. Γιατί αν έρθετε στο κέντρο φιλοξενία του Δήμου Λέσβου, που αυτή τη στιγμή έχουμε 800 ανθρώπου, φιλοξενούμε 800 ανθρώπου, έχουμε φτάσει σε αριθμό 1.800 ανθρώπων. Αυτό το κέντρο άρχισε με αριθμό 5.000 ανθρώπων. Πιστέψτε με, είμαι από την πρώτη στιγμή εκεί πέρα μέσα. Μέσα στο χωριό, μέσα στην ανοιχτή κοινότητα πλέον, mixed nationalities, όλες οι εθνικότητες, αλλά από την πρώτη μέρα διδάσκουμε το πνεύμα της αλληλεγγύης μεταξύ μας, το πνεύμα του σεβασμού, το πνεύμα της ελευθερίας και της οικογενειακής κατάστασης. Δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα, αν και υπάρχουν μερικά και πάντα θα υπάρχουν, γιατί έτσι είναι ο κόσμος, έτσι είναι ο άνθρωπος. Αλλά δεν έχουμε μεγάλα προβλήματα όσον αφορά τις διαφορές εθνικοτήτων και τις διαφορές θρησκείες. Γιορτάζ, πριν φύγω γιορτάζαμε το Ραμαζάνι. Και το γιορτάζουμε ακόμα. στι 27 Ιουλίου θα τελειώσει. Προηγουμένω γιορτάζαμε το Πάσχα. Πριν το Πάσχα είχαμε τα Χριστούγεννα διάφορες εθνικότητες, διάφορες θρησκείες που ζούμε κάτω από μία στέγη. Τη στέγη της οικογένειας, τη στέγη του σεβασμού και της αξιοπρέπειας. Όχι. Δεν είναι resort, δεν είναι η πιο λούξουρη κατάσταση σε όλη την Ευρώπη ή στην, Ελλάδα. Κάθε άλλο. Προσπαθούμε να κρατήσουμε με νύχια και με δόντια αυτό το κέντρο, διότι πλέον, ναι, μπορούμε να πούμε σε όλους τους ε, συνανθρώπους μας ότι μπορούμε να δώσουμε τη φιλοξενία μας σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη με αξιοπρέπεια. Αυτό μπορούμε να πούμε μόνο. Δεν είναι θέμα ανταγωνισμού, δεν είναι θέμα ε, ε, κάποιος διαγωνισμός ποιος θα κάνει καλύτερα και ποιος θα κάνει χειρότερα. Όχι. Είναι θέμα σχεδιασμού. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να προχωρήσουν, θέλουν να πάνε παρακάτω. Η σκέψη και η λογική τους όταν αρχίζουν το ταξίδι και τους εκμεταλλεύονται οι διάφοροι αυτοί ε, επιτίδιοι εγκληματίες για μένα σε όλο το ταξίδι από την πληροφορία μέχρι και πώς θα τους οδηγήσουν. Και γιατί είπα την πληροφορία, αυτό, αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι βρισκόμαστε στο σεμινάριο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Σε ένα σεμινάριο μέσων μαζικής ενημέρωσης. Διότι εδώ μέσα υπάρχουν πάρα πολλοί δημοσιογράφοι και όχι μόνο. Γιατί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μπορούν να διαμορφώσουν γνώμες, εικόνες και μπορώ να πω σύστημα, συστήματα. Τα μέσα μαζική ενημέρωση είναι ένας δυνατός παίχτη πάνω σε αυτό που λέγεται φιλοξενία προσφύγων και μεταναστών, πάνω σε αυτό που λέγεται μάλλον γενικά στη ζωή των ανθρώπων. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να, αναλογι... μάλλον να αναλογιστεί ο καθένα μας αν κάνει τη δουλειά αυτή που πρέπει να κάνει, αμερόληπτα και αμετάκλητα, και αν θα βοηθά με αυτό που κάνει ή σαμποτάρει. Ίσως λέω μεγάλες κουβέντες. Σε αυτά τα δύο χρόνια πείρας όμως θα μου επιτρέψετε ότι να έχω ζήσει απείρου κάλους καταστάσεις στο στυλ να έρχονται μέσα και συνημέρωσης στο χώρο του κέντρου και να προσπαθούν να βρουν το ψεγάδι. Το ψεγάδι αυτό που λέμε εμείς το κουσούρι. Αυτό που λέμε εμείς οι Έλληνες το, το κακό από λίγο κακό μέχρι μεγάλο κακό. Να το κάνουμε μεγάλο κακό. Για να δείξουμε τι. Το δράμα. Να πουλήσουμε το δράμα. Όχι, εμείς δεν πουλάμε τίποτα εκεί. Ίσα ίσα που προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας, γιατί νιώθουμε ότι προσφέρουμε υπηρεσίες και όχι, ότι, και όχι ότι δουλεύουμε, απλόχερα, μέσα από την καρδιά μας και χωρί να το υπολογίζουμε. Αλλά δεν μπορούμε να επιτρέψουμε τον, τον καθέναν να εκμεταλλεύεται αυτού του ανθρώπου και να δημιουργεί άλλου είδου καταστάσει που θα είναι κακό σε αυτού. Κοιτάξτε, μην βλέπετε το δέντρο, δέστε το δάσο. Θα είναι κακό σε αυτού που ελπίζουν, κακό στην τοπική κοινωνία, κακό γενικά σε όλη την Ευρώπη. Αν θέλουμε λοιπόν να λεγόμαστε σωστοί Ευρωπαίοι πολίτε, θα πρέπει να σεβόμαστε κάθε στιγμή και ώρα αυτό που κάνουμε και αυτό που εκπροσωπούμε και πώ το κάνουμε. Θα σα πω μια ιστορία, ε, πολύ γρήγορα, για να τελειώσω. Τελειώνω εδώ, συγγνώμη κιόλα. Έχω, κατα... Έχω καταναλώσει τον χρόνο μου. Εντάξει, μπορείτε να ολοκληρώσετε. Υπάρχουν ερωτήσει πάνω σε αυτό. Ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη. Σα Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία, ας περάσουμε στην άλλη πλευρά, στην κυρία Λάτσε. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ. θα αναρωτιέστε ποια είναι η εμπειρία της Λετωνία, ποιε είναι οι δικέ μας μαρτυρίες και ε, να σας πω πω εν μέρει έχετε δίκιο. Μέχρι το 2015 δεν είχαμε καμία ε, πρακτική πολιτική ασύλου στη χώρα μας. Είχαμε περίπου 30 ε, τη ασύλου που γίνονταν δεκτές. Όμως από το 2015 και μετά η Λετωνία συμφώνησε να υποδεχτεί έναν αριθμό προσφύγων Και μπορώ να πω ότι το σύστημα ασύλου στη χώρα μας ε, φτιάχτηκε από το τίποτα. Δημιουργήσαμε στρατηγική, δημιουργήσαμε διάφορες νέες υπηρεσίες, αντλήσαμε διδάγματα από τις βέλτιστες πρακτικές ε, στην ε, γειτονιά μας, στη Σκανδιναβία, αλλά όχι και μόνο εκεί. Υιοθετήσαμε και εμείς το σύστημα των μεντόρων, των κοινωνικών λειτουργών που βοηθούσαν ανθρώπους που είχαν φτάσει στην Λετωνία. Εξυγχρονίσαμε τα κέντρα υποδοχής, τις υπηρεσίες έβρεσης εργασίας, ε, μαθήματα γλώσσας, παιδικούς σταθμού του χώρους υποδοχής. Και μέχρι τώρα έχουμε δεχτεί το 60% του αριθμού που έχουμε συμφωνήσει, 380 δηλαδή, άνθρωποι μέχρι τώρα είναι ένα αριθμό που μπορεί να μην σα φαίνεται μεγάλο, όμω είναι αυτοί που έχουν ήδη μεταγκατασταθεί ε, και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που διέσχισαν τα ρωσικά σύνορα μόνοι του. Η υποδοχή λοιπόν είναι σε καλό δρόμο, εξελίσσεται καλώ. Υπάρχουν διάφορε πρωτοβουλίε οι οποίε είναι ε, επίσης αξιόλογες υπάρχουν μη κυβερνητικέ οργανώσεις οι οποίες προσπαθούν να μας βοηθήσουν ε, σε θέματα στέγασης, παρέχουν διερμηνία. Δυστυχώς όμως το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε είναι οι δευτερογενείς μετακινήσεις. Από τους 360 ανθρώπους που τους είχαν ανατεθεί μέντορες έχουν φύγει 313. Οι περισσότεροι πήγαν στη Γερμανία, αλλά και στη Σουηδία και τη Δανία. Και φαίνεται λοιπόν, αν ε, κάνει κανείς τις ε, μαθηματικές πράξεις, ότι μας εγκαταλείπουν όλοι. Οι λόγοι είναι πολλοί. Φυσικά και έχουμε ε, αναπτύξει διάφορες υπηρεσίες για τους πρόσφυγες, όμως η, τα μηνιαία επιδόματα είναι ελάχιστα. Είναι 100 20 ευρώ περίπου για τον πρώτο μήνα. Δεν παρέχουμε στέγαση. Έχουμε μαθήματα γλώσσας άλλα δύο φορές την εβδομάδα. Δεν είναι δηλαδή αρκετά εντατικά ή όσο εντατικά όσο θα έπρεπε. και σε ό,τι αφορά τις θέσεις απασχόλησης, οι περισσότερες ε, χρειάζονται τουλάχιστον βασικές γνώσεις της γλώσσας μας και η γλώσσα μας, όπως ξέρετε, δεν είναι καθόλου εύκολη. Υπάρχουν λοιπόν διάφορα θέματα τα οποία μας δυσκολεύουν. Επίσης, εξαιτία της ε, πολιτικής κατάστασης δεν μπορούμε να αλλάξουμε πολλά. Τα επιδόματα θα παραμείνουν χαμηλά γιατί η Λετωνία δεν είναι τόσο ανεπτυγμένη ε, χώρα και το επιχείρημα που χρησιμοποιούν για να μην αυξήσουν τα επιδόματα είναι ότι δεν μπορείς να δίνεις περισσότερα στους πρόσφυγες από ό,τι στους ε, δικούς σου πολίτες. Η στέγαση είναι ένα θέμα στη Λετωνία ακριβώς γιατί έχουν διάφορα μειονοτικά προβλήματα στη χώρα μας. Ε, η γλώσσα είναι ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στην έβρεση εργασίας και η νομοθεσία δεν προβλέπεται να αλλάξει σύντομα. Αυτά λοιπόν είναι τα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και πέραν αυτών έχουμε και διάφορα θέματα συντονισμού. Γι' αυτό και φεύγει ο κόσμος από εμά. Και έχουμε προσπαθήσει να τους παρέχουμε κάποια στήριξη, όμως ε, τονίζω πως η βοήθεια αυτή είναι εθελοντική και όσο παραμένει εθελοντική δεν μπορεί να βελτιώσει πολύ τα πράγματα. Δεν μπορούμε να μετακινήσουμε Επίση του ανθρώπους αυθαίρετα, να πούμε ότι εντάξει εμείς πήραμε 60% τη ποσόστοση που έχουμε, εντάξει μέχρι το τέλος του χρόνου θα τα έχουμε καταφέρει να τους δεχτούμε όλους. Το θέμα όμω είναι ότι όταν φεύγουν δεν μπορούμε εμεί να κάνουμε κάτι. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό τα προγράμματα μετεγκατάστασης να συνοδεύονται από κονδύλια ένταξης των προσφύγων, έτσι ώστε να παρέχεται ουσιαστική βοήθεια στους πρόσφυγες που φτάνουν στη χώρα μας, στην κοινωνία μας, έτσι ώστε να μπορούν να μάθουν τη γλώσσα με εντατικά μαθήματα, έτσι ώστε να έχουν στέγαση και αυτά, αυτές οι παροχές να μην επιβαρύνουν τον εθνικό μας περιπολογισμό. Και εδώ να πω ότι αυτές οι δευτερογενείς μετακινήσεις γίνονται προς άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Γερμανία κυρίως, και πρέπει να λαμβάνετε και αυτό υπόψη όταν θα ε, δημιουργείται αυτό το νέο σύστημα συντονισμού στην Ένωση. Τι θα γίνει δηλαδή με τους πρόσφυγες αφού φτάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά όσα είχα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα η προοπτική που μας δώσατε. Από αυτά που είπατε συμπεραίνω ότι υπάρχει ε, καταρχάς ε, μια προθυμία, υπάρχει καλή θέληση, καλωσορίζουν τους πρόσφυγες ε, στην Λετωνία, από την άλλη όμως οι πρόσφυγες δεν μένουν στη χώρα σας. Και το θέμα της συζήτησης χθες είχε να κάνει με αυτό, συζητήθηκε αυτή η περίπτωση πολλών προσφύγων που ζητούν άσυλο και θέλουν να πάνε στη Γερμανία. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω πως ε, έχει έρθει η ώρα να δώσω το λόγο στην ε, Βιόλα Βίντερστάιν έτσι ώστε να μας μιλήσει για τη δική της εμπειρία στη χώρα αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Χαίρομαι πολύ που με καλέσατε. Έρχομαι από το Βερολίνο και πρέπει να σας πω ότι αυτά που έζησα στη Γερμανία δεν αντικατοπτρίζουν την κατάσταση σε όλη την ε, χώρα. Δεν είναι ενδεικτικά της κατάστασης στη Γερμανία. Από το 2015 μέχρι φέτος, μέχρι το 2017, είδαμε υπερβολικά συνήθιστα πολλούς ε, πρόσφυγες να φτάνουν στη χώρα μας, κάτι το οποίο είχε επιπτώσεις και στις δημόσιες υπηρεσίες και στην κοινωνία, δημιούργησε μεγάλες προκλήσεις. Ανήκω σε μια ανθρωπιστική οργάνωση των Ιωαννητών. Δεν είναι ίσως τόσο γνωστή σε εσά, είναι όμως μια ανθρωπιστική οργάνωση που είναι υπό την αιγίδα του Ερυθρού Σταυρού. Συνήθως ασχολούμαστε με την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε περιπτώσεις εντός 24 ωρών ε, και προσπαθούμε να προστατεύσουμε τους αστέγους κυρίως. Μέχρι τώρα αυτά. Επίσης συνεργαζόμαστε πολύ στενά με το Υπουργείο Υγείας που είναι από τα Υπουργεία που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή στην υποδοχή των προσφύγων. Ε, τώρα, το 2015 χρειαστήκαμε πολλές ε, έκτακτες ε, υποδομές στέγασης, διότι έφτασαν πάρα πολλοί πρόσφυγες στη Γερμανία, οι οποίοι είχαν ανάγκη να κοιμηθούν κάπου, να έχουν τρία γεύματα την ημέρα. Δεν υπήρχαν ε, επίσης ε, και είχαν ανάγκη για ε, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, θέλαν γιατρούς. Δεν υπήρχαν αρκετά σπίτια, αρκετά κτίρια. Ψάξαμε να βρούμε λοιπόν άδεια κτίρια, γυμναστήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις, άδεια σχολεία. Στο Βερολίνο είχαμε και πολλά εκθεσιακά κέντρα που ήταν άδεια και μπορούσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Είχαμε και ένα αεροδρόμιο που δεν χρησιμοποιείται πια. Δυστυχώς όμως ο αριθμός των προσφύγων ήταν τόσο μεγάλος που τα πράγματα είναι πολύ στενόχωρα. Και η οργάνωσή μας προσπαθεί να κάνει ό,τι μπορεί. Προσπαθούμε να μην κρατάμε πάνω από 250 ανθρώπους ε, στον ίδιο χώρο, ακριβώς για να ε, έχουμε μια καλή εικόνα της κατάστασης, να μπορούμε να ασχοληθούμε με τον καθένα ξεχωριστά και να τους φροντίσουμε. Κύριο μέλημά μας επίσης ήταν ε, να βρούμε το συντομότερο δυνατόν ένα μέρος ε, να ε, κοιμηθούν οι πρόσφυγες όταν φτάνουν. Ζητήσαμε μάλιστα βοήθεια από διάφορες χώρες και από τον Καναδά για να μας στείλουν κρεβάτια, να μας στείλουν κινητά ντους, μεταφερόμενες τουαλέτες. Αυτό όμως που διαπιστώσαμε είναι ότι αυτές οι προσωρινές ε, εγκαταστάσεις ε, τελικά δεν ήταν και τόσο προσωρινές. Οι άνθρωποι έμεναν παραπάνω από ό,τι περιμέναμε και μετά είχαν και κάποιες πρόσθετες ανάγκες. Έπρεπε να έχουν τη δυνατότητα να μαγειρέψουν, να φτιάξουν φαγητό, να... Είναι, να μπορούν να το αποθηκεύσουν σε ψυγεία, να έχουν ένα ασφαλές μέρος να αφήσουν τα πράγματά τους, να κάνουν ένα μπάνιο, ένα ντους ε, προστατευμένο. Όμως ε, οι χώροι είναι περιορισμένοι, οι διαδικασίες ασύλου κρατούν πάρα πολύ καιρό και οι ανθρωπιστικές ε, οργανώσεις όπως η δική μας δεν μπορούν δυστυχώς να επηρεάσουν την πολιτική έτσι ώστε να επισπευθεί η κατάσταση. Προσπαθούμε όμως να βοηθήσουμε ιατρικά, με φάρμακα, με γιατρούς, να συνοδεύουμε τους πρόσφυγες σε ιατρικά ραντεβού, έτσι ώστε να απολαμβάνουν τις ίδιας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης με τους ε, Γερμανούς πολίτες. Προσπαθούμε να βρούμε θέσεις για, στους παιδικούς σταθμούς για να μπορούν να είναι τα παιδιά τους ε, σε κάποια μέρη να Προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους πρόσφυγες στην αναζήτηση στέγης και μπορώ να σας μιλήσω μόνο για το Βερολίνο, αλλά είναι μια καταστροφή. Είναι απαράδεκτα τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρει ένα μέρο να μείνει, να βρει ένα διαμέρισμα, ακριβώ γιατί ακόμα και αυτοί που, ε, που έχουν μια δουλειά δεν ε, κερδίζουν αρκετά στο να μπορούν να πληρώσουν τον νίκη. και μάλιστα μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα της ε, αίτησης ασύλου είναι πολύ, ε, περιορισμένο, πολύ περιορισμένα τα δικαιώματα που έχει κάποιος. Δεν ξέρω σε άλλες χώρες αν είναι διαφορετικά τα πράγματα, αλλά ε, στο Βερολίνο, στη Γερμανία υπάρχουν προβλήματα. Και σε ό,τι αφορά την οικογενειακή επανένωση και πάλι αντιμετωπίζουμε πάρα πολλές δυσκολίες, γιατί πολλές φορές η οικογένεια έχει χωριστεί στα δύο και ε, η μισή είναι σε μία χώρα, η άλλη μισή σε άλλη. Πολλές φορές οι διαδικασίες ασύλου κρατούν μέχρι και δύο χρόνια και μπορείτε να φανταστείτε αν που μένουν σε αυτές τις προσωρινές εγκαταστάσεις τι τραβάνε. Ε, προσπαθούμε λοιπόν να τους παρέχουμε και ψυχολογική υποστήριξη. Υπάρχει γενικό σε μία αντιμετώπιση που προσπαθούμε να είναι σφαιρική Όμως έχουμε πάρα πολλά εμπόδια, τα οποία είναι πολιτικής κυρίως φύσης και πολλές φορές πρέπει να περιμένουμε πολύ καιρό για κάποια πολιτική απόφαση, μέχρι και για μεταφράσεις μιας απόφασης στη γλώσσα ε, των προσφύγων. Θα μπορούσα να μιλήσω για μία ώρα ακόμα, αλλά νομίζω πως ε, μπορώ να σταματήσω προς το παρόν εδώ. Ευχαριστούμε πολύ. Πράγματι, εκπλήσει το σκέφτηκα την ώρα που σας άκουγα. Σε τι βαθμό δηλαδή έχουμε να κάνουμε με έκτακτες καταστάσεις. Έκτακτης ανάγκης. Σκεφτόμαστε ότι η Γερμανία είναι η σούπερ χώρα που μπορεί να αναλάβει τα πάντα. Τελικά όμως το πράγμα έχει να κάνει με ανθρώπους. Τους ανθρώπους πώς θα βοηθήσουμε και θα τους προσφέρουμε δουλειά. Ευχαριστούμε πολύ λοιπόν για την δικιά σας μαρτυρία. Και τώρα στρέφομαι στον κύριο Κόβατς, ο οποίος είναι από την Ουγγαρία. Έχετε το λόγο για να μας μιλήσετε για τις δικές σας εμπειρίες. Ευχαριστώ πολύ. Όντω, έρχομαι και εγώ από μια άλλη σούπερ χώρα, υπερχώρα. Και αυτό μετά τα χθεσινά σχόλια. Τέλο πάντων, ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία αυτή που μου δίνετε, που με προσκαλέσατε πρώτα απ' όλα και μου δίνετε την ευκαιρία να σας μεταφέρω τις εμπειρίες μου. Εγώ δουλεύω για μια μη κυβερνητική οργάνωση τα τελευταία 20 χρόνια που ονομάζεται MENEDEC. Ε, είναι καταφύγιο για την προστασία των ε, μεταναστών και για την κοινωνική του ένταξη, την κοινωνική ένταξη των ξένων που βρίσκονται στην Ουγγαρία, είτε πρόκειται για τον δυσάσυλο, είτε πρόκειται για αναγνωρισμένους πρόσφυγες, είτε πρόκειται απλώς για μετανάστες που χρειάζονται κάποια κοινωνική βοήθεια. Η εικόνα της χώρας μου όσον αφορά το προσφυγικό και το άσυλο είναι πολύ άσχημη, κάτι το οποίο είναι εν μέρη πραγματικότητα. Κοιτώντα στα νούμερα θα δούμε ότι εξακολουθούν να έρχονται τούντες άσυλο που τυχαίνουν προστασία το 2016 πάνω από 400 πήραν άσυλο, κάτι το οποίο αν δούμε τι έχει γίνει τα τελευταία 10-15 χρόνια, δεν είναι άσχημα. Πάνω από 100 πήραν φέτος άσυλο, παρόλο που η χώρα ε, θεωρείται ότι έχει το χαμηλότερο ποσοστό. Πέρυσι ήταν 10%, ε, φέτος είναι 5% από αυτούς που έχουν ε, ζητήσει άσυλο ή περιμένουν ακόμα να προχωρήσει η διαδικασία. Πάντω ο κόσμος έρχεται, φτάνει στη χώρα μας και μετά θέλει να φύγει. Δεν θέλει να μείνει. Ακόμα και αυτοί που φτάνουν με το σκεπτικό «Ε, ας δοκιμάσουμε να μείνουμε εδώ». Τελικά μπορεί να αποφασίσουν και αυτοί να φύγουν. Πρόκειται για αυτή την ομάδα. Με αυτούς δουλεύουμε εμείς. 4.000 είχαμε τελευταία ετούντες άσυλο ή άλλους που χρήζουν ε, ανθρωπιστικής βοήθειας, διεθνούς προστασίας και προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε με διάφορες δραστηριότητες για να βρουν δουλειά, ε, να μάθουν τη γλώσσα ή γενικά μαθήματα γενικής κουλτούρας. Ακούμε πολλά από τον κόσμο. Γιατί δηλαδή τελικά αποφασίζουν να μην θέλουν να μείνουν στην Ουγγαρία. Ο πρώτος λόγος είναι ότι έτσι κι αλλιώς μπαίνοντα στη χώρα έχουν από πριν την πρόθεση να φύγουν να πάνε αλλού. Και ακόμα και αν μείνουν στην Ουγγαρία και να περιμένουν όλη την διεξαγωγή της διαδικασίας για το άσυλο, μπορεί να αλλάξουν γνώμη καθοδόν. Άλλοι κοιτούν γύρω τους, ακούν ότι υπάρχουν καλύτερες ευκαιρίες αλλού, στη Δυτική Ευρώπη. Και είναι ενδιαφέρον ότι ακριβώς το χαμηλό ποσοστό αναγνώρισης δεν είναι ο κύριος λόγος. Δεν μοιάζει τον κόσμο τόσο πολύ το ποσοστό αναγνώρισης ασύλου. Έτσι κι αλλιώς πιστεύουν ότι ο λόγος για τον οποίο έχουν βρεθεί και που έχουν βρεθεί είναι απόλυτα θεμητό. Η Ουγγαρία λοιπόν έχει πολύ καλή φήμη όσον αφορά την πολιτική της για αυτό το θέμα. Πολλές λοιπόν ε, οι οικογένειες θέλουν να φύγουν, να πάνε στη Γερμανία, τη Σουηδία, τις κατοχώρες και πιστεύουν, ελπίζουν ότι εκεί θα είναι πιο εύκολο να καταφέρουν να καταλήξουν σε επανένωση με τις οικογένειές τους. Και έπειτα υπάρχουν και τα κοινωνικά ωφέλη που κάνουν τον κόσμο να φύγει από τη χώρα. Γιατί και εδώ η Ουγγαρία δεν προσφέρει πολλά. Πέρυσι, μετά από ένα συνολικό πακέτο περιορισμού του συστήματος ασύλου, έκοψε τη κοινωνική στήριξη στους πρόσφυγες ή σε αυτούς που χαίρουν επικουρικής βοήθειας. Και δεν υπάρχει επίσημη στήριξη λοιπόν για αυτούς οι οποίοι αναγνωρίζονται όσο χρήζονται σε ανθρωπιστική βοήθεια. Πρόκειται περισσότερο για κονδύλια που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το ΑΜΙΦ, που πάνε στην κυβέρνηση και η κυβέρνηση έτσι κι αλλιώς συνεισφέρει σε αυτό το Ταμείο. Αλλά πρόκειται, όπως καταλαβαίνετε, για πολύ περιορισμένους πόρους. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι πάρα πολλές. Πρώτα απ' όλα η στέγαση πώς να βρεθεί στέγαση για τους ανθρώπους αυτούς. Όσοι φεύγουν από το σύστημα ασύλου υποδοχής, πηγαίνουν τελικά σε ένα καταφύγιο για άστεγους. Που τα καταφύγια αυτά οργανώνονται από, μέσω κονδυλίων από το ΜΙΦ. Δεν είναι αδύνατο να βρει κανείς δουλειά, αλλά σίγουρα είναι πολύ δύσκολο. Οι άνθρωποι καταλήγουν στην εθνική οικονομία. Ε, χτες ακούσαμε ότι μερικές φορές αυτό μπορεί να είναι θετικό, αλλά τις περισσότερες φορές τους εκμεταλλεύονται. Γιατί δουλεύουν αυτοί οι άνθρωποι για δύο ευρώ την ώρα. Από εκεί ξεκινάνε και καταλαβαίνετε ότι δεν φτάνουν. Και το τελευταίο είναι η εχθρική στάση του κόσμου, αλλά και του κράτους. Αν ακούσει κανείς τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, δεν κάνουν καμία διάκριση ανάμεσα σε αυτούς που χρειάζονται ανθρωπιστική προστασία και τους υπόλοιπους. Δεν γίνεται αυτή η διάκριση. Οπότε η ρητορική οδηγεί στο να υπάρχουν όλο και λιγότερες ευκαιρίες για ένταξη των ανθρώπων αυτών στις τοπικές κοινωνίες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κόβατς, πολύ ειλικρινή όσα μας είπατε. Το κοινό που βλέπω εγώ από όλα όσα άκουσα μέχρι τώρα, σήμερα, είναι το θέμα της επανένωσης των οικογενειών. Φαίνεται ότι είναι κάτι πολύ ζωτικό όσον αφορά την πολιτική ασύλου, γιατί τελικά μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι ψάχνουν μια καινούρια ζωή, όχι μόνο για τους αυτούς τους ως άτομα, αλλά για τις οικογένειές τους επίσης. Πολύ ενδιαφέρον παράγον αυτός. Βέβαια, Αυτά που είπατε μου θυμίζουν και αυτά που ακούσαμε χτες από την Σόφη Μακέλης, η οποία είπε ότι όταν τα μέσα ενημέρωσης αναφέρονται σε τούτες άσυλο μετανάστες και πρόσφυγες, έχει σημασία η γλώσσα που χρησιμοποιούν. Και βλέπουμε και εδώ το αρνητικό παράδειγμα ότι ακόμα και ο δημόσιος λόγος προκαλεί σύγχυση, μάλλον επίτηδες, μπερδεύει τις διαφορές έννοιες. Σας ευχαριστούμε πολύ λοιπόν για αυτά. Τελευταίος. Η τελευταία μαρτυρία είναι από τον κύριο Πιέρ Φαρμπέρεν, ο οποίος είναι Βέλγος και είναι Γενικός Διευθυντής της Οργάνωσης Γιατρών του Κόσμου Βελγίου. Σίγουρα θα μας πείτε κι εσείς ποια είναι η εμπειρία σας στο Βέλγιο και περί τίνος πρόκειτο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για την πρωτοβουλία αυτή και σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε εδώ σήμερα. Πράγματι, όπως ακούσαμε και πριν, είναι η δίγηση, ο τρόπος που αναφερόμαστε σε αυτά τα θέματα, φτιάχνει συνειδήσεις και είναι προφανές ότι στο διάλογο αυτό, με αυτούς οι οποίοι φτιάχνουν συνειδήσεις, πρέπει να είναι προτεραιότητα για μας. 2.000 άνθρωποι κάθε μέρα πάνε στην Ουγκάντα φεύγοντας από το νότιο Σουδάν. Όπως το ίδιο νούμερο όπως στη Γερμανία το 2015. Πρόκειται για τις ίδιες δουλειές και η Ουγκάντα αποφάσισε να αναθέσει δύο εκτάρια στο καθένα για να μπορέσει να ζήσει αξιοπρεπώς. Είναι και αυτός λοιπόν ένας τρόπος εντελώς νέος υποδοχής ε, προσφύγων. Είναι πολύ ενδιαφέρον να σκεφτούμε πρώτα τη ζωή πριν περάσουμε στα διοικητικά, την καταγραφή που αποτελούν ουσιαστικά και την δισκαμψία της Ευρώπης να δει πρώτα τον άνθρωπο πριν δει τους διοικητικούς κανόνες που πρέπει να ακολουθήσει αυτός για να μπορέσει να ζήσει. Έτσι λοιπόν, εμείς είμαστε παρόντες 110 πόλεις στην Ευρώπη για να συνοδεύσουμε τους μετανάστες δεν είμαστε μόνο εκεί που υπάρχει κρίση, Λέσβος φυσικά, Καλαβρία και το Καλέ, Grand Σαντ, ε, αναφέρθηκε σε αυτά ο Καρέν πριν από λίγο. Είμαστε παρόντες όμως και σε άλλες πόλεις, στην καθημερινότητα των μεταναστών και όταν δουλεύουμε με τους μετανάστες, αυτό το οποίο είναι πιο σημαντικό για μας είναι ότι αναγκαζόμαστε να καλύψουμε μία κατάσταση που καλύπτουν άνθρωποι που δεν είναι υπεύθυνοι για αυτά. Γινόμαστε ειδικοί χρησιμοποιώντας την νομοθεσία έτσι ώστε κάθε φραγμό στην πρόσβαση, στη στέγαση, στην απασχόληση, στην υγεία κτλ. να πάψει να υπάρχει, να καταργηθεί. Όμως τα εμπόδια αυτά είναι πάρα πολλά και γι' αυτό αυτό φτιάχνουν την καθημερινότητα των μεταναστών οι οποίοι τελικά δεν μπορούν να δουλέψουν αν δεν έχουν περιμένει προηγουμένω του χώρου υποδοχή για μήνε και μήνε. Αυτή είναι η καθημερινότητα των ε, προσφύγων, οι οποίοι πρέπει πρώτα να καταγραφούν στι κοινωνικέ υπηρεσίε, ενώ όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν ένα σχέδιο στο μυαλό τους και το σχέδιό τους είναι να συνεισφέρουν, να συμμετάσχουν στην καθημερινότητα. Αν ε, δείτε λοιπόν τι γίνεται στα κέντρα υποδοχής για τους ετούντες άσυλο, δεν μπορούν να μαγειρέψουν. Το είπατε και εσείς πριν και σας ευχαριστώ που το επισημάνατε. Δεν μπορούν να εργαστούν. Άρα έχουμε να κάνουμε με μία μεταχείριση που τους αντιμετωπίζει σαν ε, άρρωστους, σαν ε, κακούς. Συνεπώς πρέπει να φροντίσουμε οι άνθρωποι αυτοί να μπορέσουν να ζήσουν φυσιολογικά οι ειδικοί σε θέματα υγείας λένε ότι 85% των παραγόντων που καθορίζουν την υγεία δεν είναι ιατρικής φύση. Οι άνθρωποι είναι καλά στην υγεία του επειδή ζουν κανονικά. Έχουν μια δουλειά, στέγαση κτλ. Όχι επειδή είναι καλό το σύστημα υγείας εκεί που ζουν. Αυτό ισχύει μόνο για το 15% των περιπτώσεων. Και αν πάρουμε και τι στατιστικέ των ε, γιατρών του κόσμου, από τους χίλιους που έχουμε συναντήσει, που έχουν υποστεί βία μέχρι να φτάσουν, το 57% λένε ότι είναι σε πολύ καλή υγεία. Συνεπώς το πρόβλημα, παρά το γεγονός ότι πέρασαν από βίες καταστάσεις, δεν είναι πρόβλημα υγείας. Φυσικά και υπάρχουν κάποια προβλήματα υγείας, αλλά το πρόβλημα δεν είναι υγεία. Το κύριο πρόβλημα είναι η συνέπεια της δικιάς μας μεταναστευτικής πολιτικής, η συνέπεια της διαδρομής που ακολούθησαν οι άνθρωποι αυτοί και η συνέπεια της δυσκολίας ένταξης και δυσκολίας συμμετοχής των ανθρώπων αυτών. Αυτό είναι που έχει φοβερά αρνητικέ συνέπειες επί της υγείας τους. Συνεπώς βρισκόμαστε και πάλι με δύο κατηγορίες δυσκολίας. Η μία είναι ε, ψυχικοί που δυσκολεύονται να κοιμηθούν, έχουν αυτοκτονικές τάσεις, κατάθλιψη. Γιατί είτε κατά τη διαδρομή μέχρι να φτάσουν σε εμά, είτε στην καθημερινότητά τους, περιμένοντας αποφάσεις, περιμένοντας δυνατότητες ένταξης, οι άνθρωποι αυτοί ζουν πάρα πολύ δύσκολα, οπότε υπάρχουν προβλήματα ψυχικής υγείας που είναι πάρα πολύ σημαντικά για τους μετανάστες και από την άλλη μεριά η άλλη κατηγορία προβλήματος είναι τα όσα πέρασαν στην ε, διαδρομή μέχρι να φτάσουν σε μας στην Καλαβρία. Για παράδειγμα, έχουμε 200 περιπτώσεις. που μας ε, έρχονται από τη Λιβύη αλλού, επειδή ακριβώ εκεί ήταν πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Για να αντιμετωπίσουμε λοιπόν τα προβλήματα αυτά πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τα θέματα της ψυχικής υγείας και τα άλλα. Κυρίως όμως το θέμα της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας. Αυτό λοιπόν που πάντα λέμε και κάνουμε είναι ότι δεν πρέπει τους μετανάστες να τους εντάξουμε σε ένα διαφορετικό σύστημα υγείας από το κανονικό, από το γενικό. Το να φτιάξουμε επικουρικές ε, υπηρεσίες υγείας σημαίνει ότι δημιουργούμε πάντα εμπόδια στην πρόσβαση στην υγεία. Κοστίζει ακριβά, δημιουργεί προβλήματα ε, στο κανονικό σύστημα υγείας, διακρίσεις, διακρίσεις σε βάρος του πληθυσμού υποδοχής στην Ελλάδα, για παράδειγμα. Και εδώ ο συνάδελφος σίγουρα μπορεί να σας τα πει φυσικά καλύτερα από μένα. Στην Ελλάδα λοιπόν κάποιοι καταβλισμοί προσφύγων προσφέρουν ε, συνθήκες πρόσβασης στην υγεία πολύ καλύτερες από ό,τι έχει ο ντόπιος πληθυσμός. Αυτά τα συστήματα λοιπόν τα επικουρικά οδηγούν σε διακρίσεις, οδηγούν σε προβλήματα αποτελεσματικότητας και δημόσιας υγείας. Συνεπώς, η καλή πρακτική είναι οικουμενικής, καθολικής κάλυψης, όπου και οι μετανάστες θα έχουν την ίδια πρόσβαση στην υγεία όπως και ο ντόπιος πληθυσμός. Και είναι αυτές οι πρακτικές που επιτρέπουν και στον κόσμο να φέρουν τις μαρτυρίες τους, τις ε, εμπειρίες τους από τη διαδρομή που ακολούθησαν και να μιλήσουν και για τα σχέδιά τους. Να βγούνε ίσως από τις δικές μας δομές. Εμείς έχουμε μια λογική φύλαξης του κόσμου. Όμως οι άνθρωποι πρέπει να μπορούν να ελέγχουν και τις προπτικές τους και την υγεία τους. Να τους βοηθήσουμε λοιπόν, έχουν πρόσβαση στη νέα τεχνολογία τις νέες τεχνολογίες έτσι ώστε να μπορέσουν να υλοποιήσουν τα σχέδια με τα οποία μας έφτασαν, να χρησιμοποιήσουν το κεφάλαιο που διαθέτουν. Όσοι λοιπόν ε, χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες ή τις έχουν, έχουν δημιουργήσει κάποιες εφαρμογές μπορούν να βοηθήσουν ακόμα περισσότερο τους μετανάστες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Τι βλέπουμε από αυτά που ακούω ότι είναι συστημικό ζήτημα. Και κάνουμε εξαιρετισμό με αυτά που συζητήσαμε και χτες στο θέμα της πολιτικής και το συνδέουμε με το σημερινό. Και λέμε ότι είναι σημαντικό ένα κοινό σύστημα ασύλου, αλλά δεν αποτελεί πανάκια, δεν λύνει τα προβλήματα. Είναι το θέμα προσβάσεως στην υγεία, πρέπει να βοηθήσουμε τον κόσμο να ζήσει τη ζωή του και να ξαναβρει τη ζωή του που διακόπηκε να μπορούν να μαγειρεύσουν, να δουλέψουν, να μπορούν να στηριχθούν αυτοί και τα μέλη της οικογένειάς τους. Βασικά θέματα. Άρα μιλάμε για ανθρώπους. Δεν μιλάμε για κάτι αφηρημένο. Θα διακόψουμε εδώ τις εργασίες του πάνελ. Και αυτό διότι αναμένεται η άφηξη του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του κυρίου Αντώνιο Ταγιάννη, που θα ήθελε να μας μιλήσει για ένα κοσάλεπτο μισή ωρίτσα. Ίσως μπορούμε να συνεχίσουμε τις εργασίες του πάνελ μετά, σύντομα, 10 λεπτά, ένα τέταρτο, διότι είναι σημαντικό να υπάρξει διάλογος. Λοιπόν, σας ευχαριστώ για μια ακόμη φορά. Σας ευχαριστώ για τις μαρτυρίες που παρουσιάσατε. Νομίζω ότι πράγματι δώσατε μια άλλη διάσταση, διαφορετική διάσταση, σε αυτά που συζητούσαμε χθες. Σας ευχαριστώ. Υπότιτλοι Ευχαριστώ. Ε, buenos Καλή σας μέρα. Και σας ευχαριστώ πολύ που είσαστε εδώ. Στα ισπανικά θα σας μιλήσω εγώ. Οπότε βάλτε τα ακουστικά σας για να μπορείτε και να με καταλάβετε. Να είναι πιο εύκολο έτσι να επικοινωνήσετε και με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον κύριο Αντώνιο Ταγιάννη, ο οποίος ε, δέχτηκε ε, μεγάλη χαρά να έρθει και να συμμετάσχει στο σεμινάριο αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ λοιπόν που θελήσατε να έρθετε δύο μέρες, να περάσετε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να εξετάσετε, να συζητήσετε με τους ευρωβουλευτές και τους διάφορους παράγοντες που ασχολούνται με την μετανάστευση και κυρίως με το ζήτημα του ασύλου για τους πρόσφυγες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος νομίζω για να ολοκληρωθεί το σεμινάριο αυτό από το να έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να δούμε τι έχει να μας πει και εφόσον υπάρχει χρόνος να απαντήσει και στις ερωτήσεις σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε. Ευχαριστώ σας. Καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για μένα είναι μεγάλη χαρά να μιλώ με τους δημοσιογράφους. Αφιέρωσα 20 χρόνια τη ζωής μου κάνοντας τη δουλειά σας. Και πιστεύω ότι ο ρόλος σας είναι σημαντικός για να εξηγείτε στους ε, πολίτες τι κάνουμε, σαν θεσμικά όργανα της Ευρώπης για να δώσουμε απαντήσεις στα προβλήματα των πολιτών. Το θέμα του ασύλου, το θέμα της μετανάστευσης μαζί με το ζήτημα της καταπολεμήσεως της τρομοκρατίας και της καταπολεμήσεως της ανεργίας των νέων αντιπροσωπεύουν όλα αυτά προτεραιότητα για όλους μας. Εξάλλου, αυτό εγγράφηκε στο έγγραφο που υπογράψαμε στις 25 Μαρτίου στη Ρώμη επί τη ευκαιρία της 60ης επαιτίου της υπογραφής των συνθήκων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δεσμευθεί και είναι στην πρώτη γραμμή πάνω σε αυτό στο να δώσει συμβολή αποφασιστική όσον αφορά την επίλυση του προβλήματος. Οι πολίτες ζητούν απαντήσεις ταχείες και συγκεκριμένες. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στους αυτούς μας να χάσουμε κι άλλο χρόνο, εάν δεν θέλουμε να χάσουμε την αξιοπιστία μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, όλα και τα τρία θεσμικά όργανα μαζί με τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εκτελέσουν το καθήκον τους. Πρέπει να επιταχύνουν ε, την εξέβρεση λύση των προβλημάτων. Εμείς, κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνόδου της Ολομελίας στο Στρασβούργο, εγκρίναμε ένα έγγραφο με πολύ μεγάλη πλειοψηφία και στο έγγραφο αυτό ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δράσει προς επίλυση του προβλήματος της κατανομής των προσφύγων εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Υπάρχει συμφωνία που ελήφθη στο Συμβούλιο από πλευράς κρατών μελών και τα κράτη-μέλη έχουν υποχρέωση να εκτελέσουν, να συμμορφωθούν με τη συμφωνία. Ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρέμβει και να καταστήσει σεβαστή αυτή τη συμφωνία ακόμα και μέσω διαδικασίας κατά παράβαση έναντι των κρατών εκείνων που δεν σέβονται τις ε, ληφθείσες αποφάσεις. Και για εκείνες ισχύει η αρχή ότι θα πρέπει να τηρηθούν συμφωνίες. Pacta sum servanta. Από αυτή την έποψη η θέση του Κοινοβουλίου είναι σαφέστατη. Υπάρχει τεράστιος αριθμός προσφύγων που είναι στην Ιταλία, είναι στην Ελλάδα. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να λυθεί. Πρέπει να λυθεί επίσης και αυτό συζητούμε. Χθε συναντήσατε μάλιστα τους διάφορους εισηγητές που για το πακέτο της μεταρρύθμισης του Διβλίνου πρέπει να λυθεί, λέω, και το πρόβλημα του ασύλου. Εμείς ε, θα πρέπει στην Ευρώπη να έχουμε κανόνες, κοινού κανόνες, που πρέπει να εφαρμόζονται παρομοίως παντού. Σήμερα οι κανόνες δεν είναι αποτελεσματικά εναρμονισμένη. Να σας δώσω ένα παράδειγμα που δείχνει ότι πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα. Εδώ και κάποιες εβδομάδες πήγα επίσκεψη σε δύο πόλεις μεθοριακές που είναι και σύμβολο του διαλόγου εντός Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Γκορίτσια και μια άλλη πόλη στην Σλοβενία πριν ήταν μια πόλη χωρισμένη στα δύο και τώρα είναι δύο πόλεις ξεχωριστές ε, που έχουν το κοινό στόχο στα σύνορα. Λοιπόν, στους δρόμους της πόλης, κυρίως στην Κορίτσια, υπάρχουν εκείνοι που ζητούν άσυλο, που ελπίζουν να αποκτήσουν άσυλο από την Ιταλία, έχοντας απορριφθεί αίτησή τους στην Αυστρία και στη Γερμανία. Αυτό συμβαίνει διότι δεν υπάρχουν οι ίδιοι κανόνες, δεν υπάρχει ο ίδιος κατάλογος για κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Υπάρχουν χώρες που θεωρούνται χώρες κινδύνου και αλλού δεν θεωρούνται. Το Αφγανιστάν σε κάποιες, κάποιες περιοχές του Αφγανιστάν για κάποιες χώρες θεωρούνται επικίνδυνες περιοχές, άρα δίνεται άλυσο για αυτούς που έρχονται από εκεί. Για άλλες χώρες δεν είναι επικίνδυνες περιοχές, άρα δεν υπάρχει υπόθεση για να δοθεί άσυλο. Εμείς δεν μπορούμε να έχουμε ανθρώπους που τριγυρνάνε σε όλη την Ευρώπη προσπαθώντας να βρουν άσυλο. Θα πρέπει ο κανόνας να είναι κοινό για όλους. Αν ισχύει το άσυλο στη Γερμανία πρέπει να ισχύει στην Ιταλία. Δεν ισχύει στην Ιταλία. Στη Γερμανία δεν μπορεί να ισχύει στην Ιταλία. Δεν ισχύει στην Ελλάδα, δεν πρέπει να ισχύει στην ε, Αυστρία. Αν δεν ισχύει στο Λουξεμβούργο, δεν μπορεί να ισχύει στη Μάλτα. Διαφορετικά θα έχουμε shopping, θα ψωνίζει ο άλλος άσυλο. Ο πρόσφυγας θα πρέπει εμείς να, για να έχουμε αξιοπιστία να δίνουμε το άσυλο σε εκείνον που δικαιούται ασύλου διότι προέρχεται από μια περιοχή όπου είναι επικίνδυνο να μείνει και να ζει κανείς. Παραμονές λοιπόν του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τέλους του μηνός θα οργανώσουμε σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μία διάσκεψη υψηλού επίπεδου με θέμα τη μετανάστευση. Θα γίνει στις 21 του μηνός και θα προσπαθήσουμε να συζητήσουμε το θέμα της μετανάστευσης και το δικαίωμα του ασύλου μαζί. Όλα όσα αφορούν το μεταναστευτικό φαινόμενο για να ούτως ώστε στις 22 και 23 να πιέσουμε το Συμβούλιο να υιοθετήσει αποφάσεις που θα ακολουθήσουν την κατεύθυνση γρήγορης λύσεως των προβλημάτων. Εμείς θα καλέσουμε όχι μόνο πολιτικούς, αλλά και μη κυβερνητικές οργανώσεις, εκείνους που βοηθούν τους μετανάστες στη θάλασσα, τους διασώστες, εκπροσώπους ε, της Αφρικής. Θα καλέσουμε διάφορες προσωπικότητες που μπορούν να αντιμετωπίσουν μαζί και να συζητήσουν το πρόβλημα. Σας λέω αμέσως ότι το Κοινοβούλιο εργάζεται, προσπαθεί να εγκρίνει την πρόταση του Επιτρόπου Μίμητσα για επενδύσεις στην Αφρική. Θα πρέπει να δούμε τι θα συμβεί στην Αφρική τα επόμενα 10-20 χρόνια. Υπάρχει ένα πρόβλημα που αφορά την αλλαγή του κλίματος. Ε, ε, όπου η έρημος επεκτείνεται, η Σαχάρα εκτείνεται και συνεχώς καταστρέφει καλλιεργούμενες γεές. Οπότε εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την περιοχή τους. Μπόκο Χαράμ που σπέρνει τον τρόμο μεταξύ μουσουλμάνων, χριστιανών, απάγει, σκοτώνει, καταστρέφει. Υπάρχει αστάθεια σε πολλές χώρες. Και στο Κονγκό Υπάρχουν προβλήματα στον Ήγυρα. Στην ακτή Ελεφαντοστού, στην Ιγυρία. Ε, τι συμβαίνει στη Σομαλία. Πέρα από τις μάχες μεταξύ των διαφόρων ομάδων, πέρα από την ύπαρξη των τρομοκρατών, υπάρχει και, ε, και η πείνα που, που σκοτώνει χιλιάδες παιδιά που δεν μπορούν να επιβιώσουν. Και όπως είπε και ο πρόεδρος της Αφρικανικής Ενώσεως που καλέσαμε στη συνεδρίαση, στην Ολομέλεια, σαν φιλοξενούμενο, τιμούμενο φιλοξενούμενο, μας είπε λοιπόν ότι όταν χάνεται η ελπίδα, γυναίκες και άντρες παίρνουν τα παιδιά τους παίρνουν τα λίγα υπάρχοντά τους και εγκαταλείπουν το σπίτι τους. Στην Αφρική συμβαίνει αυτό. Εκατομμύρια άνθρωποι κινδυνεύουν να χάσουν την ελπίδα. Εκατομμύρια άνθρωποι θα προσπαθήσουν να μετακινηθούν από τα νότια μέρη του κόσμου προς τα βόρεια, περνώντας τη Λιβική έρημο και διασχίζοντας τη Μεσόγειο. Αυτό σημαίνει ότι αν δεν υπάρξει μια σοβαρή στρατηγική με επενδύσεις μεγάλες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, θα έχουμε ακόμα νεκρούς στην έρημο, νεκρούς στη Μεσόγειο και θα έχουμε εκατομμύρια ανθρώπους που θα κοιτάνε προς την Ευρώπη, θα θέλουν να έρθουν προς την Ευρώπη. Μετά θα είναι δύσκολο να τους υποδεχθούμε και να τους εντάξουμε. Καλέσαμε τον Κοινωνικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για να μιλήσει για αυτό στην επόμενη σύνοδο. Ο, ο πρόεδρος Ακτής Ελεφαντοστού θα έρθει για να μιλήσει για το πρόβλημα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δηλαδή εκτελεί το καθήκον του, προσπαθεί να αντιμετωπίσει ένα θέμα το οποίο είναι στην καρδιά των πολιτών και στην καρδιά των Αφρικανών. Θέλουμε να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα με τη συμμετοχή και των Αφρικανών. Και θα συνεχίσουμε να εργαζόμεθα προς αυτή την κατεύθυνση. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι είναι σωστό ε, να έχουμε και πεδία υποδοχής και στα νότια της Σαχάρας, κέντρα υποδοχής, όπου θα υπάρχουν τρόφιμα για άντρες και γυναίκες και τρόφιμα ειδικά για τα παιδιά. Θα υπάρχουν γιατροί, να υπάρχουν νοσοκομεία εκστρατείας και να προστατεύονται και από τους ε, διακινητές και τους εμπόρους ανθρώπων που δεν ξέρουν σύνορα αυτοί και όρια. Αυτοί οι κύριοι κερδοσκοπούν από το μαρτύριο και τα βασανιστήρια του άλλου. Θα πρέπει η Ευρώπη να παίξει ένα ρόλο μέσω πολιτικής ασφαλείας τέτοιων που να εγγυάται την ε, ελευθερία αυτών των ανθρώπων. Ούτω ώστε για να γίνει αυτό χρειάζονται δισεκατομμύρια ευρώ αλλά ε, χρειάζεται και μια μεγάλη συμμετοχή ε, των εθνών που θα είναι και των Ιτιουργία, συγγνώμη. Γι' αυτό καλέσαμε να μιλήσει και να συζητήσει μαζί μας ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο κύριος Γκουτιέρες, που όχι μόνο έκανε μια, να μην κάνει μόνο μια ομιλία στο Στρασβούργο, δεν έκανε μόνο αυτό, αλλά συμμετείχε και στη διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλευτικών Ομάδων. Θέλουμε να το κάνει αυτό για να γίνει μια ανταλλαγή απόψεων τι, σκε, τι σκέφτεται να κάνει ο ΙΕ, τι σκέφτεται να κάνει, τι κάνει και πώς μπορούμε να συνεργαστούμε καλύτερα μεταξύ μας, εμείς με τον ΟΗΕ. Το Κοινοβούλιο θέλει να παίξει ένα ρόλο πρωταγωνιστικό για να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις στις απαιτήσεις που δημιουργούνται όσον αφορά τα, άτομα, τους Ευρωπαίους πολίτες και τις ανάγκες των Αφρικανών, να λάβουμε υπόψη, που είναι και θα είναι υποχρεωμένοι να εγκαταλείψουν ε, τα σπίτια τους διαφορετικά. Είναι μεγάλη πρόκληση αυτή. Δεν μπορεί να λυθεί μόνο από μια χώρα μπορεί να λυθεί μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο, ο πρόεδρος Επιτροπής της Αφρικανικής Ενώσεως και όσον αφορά τη Λιβύη ε, ζήτησε από μας να φροντίσουμε να υπάρξει μόνο ένας Ευρωπαίος ομιλητής και συνομιλητής για την επίλυση του προβλήματος στη Λιβύη πρέπει η Ευρώπη να δράσει ενωμένη. Να μην υπάρχουν πολλοί συνομιλητές που να μιλάνε με άλλους αντίστοιχους ε, συνομιλητές Λίβιους διότι η Λιβύη περνά στιγμές πολύ δύσκολες, δεν έχει σταθεροποιηθεί ακόμα και εμείς οι Ευρωπαίοι ε, μας ζητούν από εμάς Ευρωπαίους να μιλήσουμε με μία φωνή. Αυτό θέλει να κάνει το Ευρωκοινοβούλιο. Αυτό προτίθεται να στηρίξει. Θα το υποστηρίξω και εγώ στη δική μου παρέμβαση, στο επόμενο Συμβούλιο, στην ομιλία μου. Θα πάω στο Συμβούλιο ισχυρός λόγω της υποστήριξης που θα τύχω μετά από μια ημερίδα εργασιών που θα αφιερώσει το Ευρωκοινοβούλιο στο θέμα μετανάστευση. Εκεί πρέπει να ακουστεί δυνάτη η φωνή του μόνο εκλεγμένου θεσμικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που θα απευθυνθεί προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στους προσώπους των κρατών μελών. Λίγο πολύ αυτό είναι το πολιτικό πλαίσιο εντός του οποίου κινούμαστε. Αυτές είναι οι πολιτικές προτεραιότητες του Κοινοβουλίου. Ακούσατε τους εισηγητές χθες πιθανότατα που θα αναφέρθηκαν πάνω στα ζητήματα τεχνικής φύσεως. Η συζήτηση συνεχίζεται, αλλά εμείς επαναλαμβάνω, θα κάνουμε αυτό που μας αρμόζει και όπως υποσχέθηκα την ημέρα που υπογράφηκε το έγγραφο της Ρώμης, θα επαγρυπνεί το Κοινοβούλιο το ώστε οι δεσμεύσεις των θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών θα γίνουν σεβαστές και θα εφαρμοστούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ακουστούν κάποιες ερωτήσεις, αν θέλετε, πριν ε, φύγει ο Πρόεδρος. Είσαστε προσκεκλημένοι βέβαια για αυτήν την υψηλού επίπεδου διάσκεψη και ε, ο Μασιμό θα σας ενημερώσει περισσότερο στο τέλος της συζήτησης. Παρακαλώ για ερωτήσεις. Εσείς. Uh, my name is uh, Ονομάζομαι Ούτ, δημοσιογράφος από την Blood της Σουηδίας. Θα ήθελα να σας ζητήσω να μου πείτε δύο λόγια για την επικοινωνία που έχετε με την Λιβύη. Πώς θεωρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θα είναι η συμφωνία με την Λιβυκή πλευρά. Συνεργαζόμαστε με την κυβέρνηση στην Τρίπολη. Υποδέχθηκα μάλιστα και τον ε, νέο αρχηγό της κυβέρνησης της Βρυξέλλες. Υπάρχει μια συμφωνία ανάμεσα στην Ιταλία και τη Λιβύη, την οποία στηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. έτσι ώστε να σταματήσει η παράτυπη μετανάστευση. Υπάρχουν Ιταλικές και Ευρωπαϊκές επενδύσεις που στηρίζουν αυτή τη συμφωνία, που στηρίζουν την ε, ακτοφυλακή της Λιβύης. Δυστυχώς όμως η κατάσταση στη Λιβύη είναι περίπλοκη. Υπάρχουν πολλά προβλήματα και στην κυβέρνηση, στην Τρίπολη, αλλά και αλλού, και στο Τομπρούκ, όπως γνωρίζετε. Στη Λιβύη είναι σαν να υπάρχουν δύο χώρες σε μία. Κυριναϊκή και Τρίπολη. Είναι χωρισμένη η χώρα στα δύο. Ο βασιλιάς Ίντρης το 1960 πήγε στο Τομπρούκ και ο Καντάφη, ο ηγέτης της Πράσινης Επανάστασης, γεννήθηκε στην Τρίπολη, κοντά στην Τρίπολη. Και η πρώτη επίθεση εναντίον του Καντάφη έγινε από την Κυριναϊκή. Υπάρχουν όμως και πολλά προβλήματα στο Νότο. Υπάρχουν ε, οι μουσουλμανοί αδελφοί υπάρχουν μάχες. Είναι γι' αυτό λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει ένας συνομιλητής τον οποίο θα στηρίζουμε και ο οποίος θα στρώσει το δρόμο για την επανένωση της χώρας. Είναι λοιπόν δύσκολα τα πράγματα εκεί. Πρέπει όμως να προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε με τους ε, Λιβύους έτσι ώστε να έχουμε μία λύση που θα είναι τόσο για εμάς καλή όσο και για όσους ε, έρχονται από τα νότια. Ναι, ε, να ρωτήσω και κάτι επιπλέον. Πώς μπορείτε να έχετε εμπιστοσύνη στους συνομιλητές σας. Πώς μπορείτε να εμπιστεύεστε κάποιον που προέρχεται από ε, μια διαλυμένη χώρα όπως η Λιβύη. Απάντηση. Πρέπει να στηρίξουμε μία κυβέρνηση μόνο. Να επιλέξουμε. Δεν είναι εύκολο αυτό αλλά πρέπει να επιλέξουμε μία και να τη στηρίξουμε και σε τεχνικό επίπεδο, να προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε με την κυβέρνηση αυτή. Αλλά και για την πολιτική ασφαλείας πρέπει να ενισχύσουμε το στρατό, την ακτοφυλακή τους, γιατί χρειάζεται δημοκρατία και η δημοκρατία δεν είναι εύκολο πράγμα. Πρέπει όμως να προσπαθήσουμε να σταθεροποιήσουμε τα πράγματα και αυτή Μία τελευταία ότι θα είναι η μόνη λύση. Μία τελευταία ερώτηση θα δεχτούμε. Εσείς παρακαλώ. Κοιτάξτε. Λοιπόν, μοιρασμό των ευθυνών είναι μια τελευταια ερωτηση θα δεχτουμε εσει παρακαλω κοιταξτε λοιπον μοιρασμο των ευθυνων ειναι μια εννοια του Δουβλίνου, έτσι. Επιμοιρασμό. Τι, τι κάνουμε με του τέσσερι του Βίζογκραντ. Δεν ξέρω αν συμφωνεί ο Βίκτορ Ορμπάν. Αναφερθήκανε κάποιε κυρώσει. Τι θα συμβεί με αυτή την ιστορία. Πρόεδρο, εγώ μίλησα για το σεβασμό των ευρωπαϊκών κανόνων. Υπάρχει μια συμφωνία που επετεύθη σε επίπεδο Συμβουλίου. Αν δεν γίνει σεβαστή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία επί παραβάση έναντι των χωρών που δεν σέβονται τη συμφωνία. Δεν είναι κάτι εναντίον του μυαλού ή του άλλου. Είναι θέμα συμφωνία. Ισχύει για όλου. Η διαδικασία κατά παράβαση είναι, ξεκινάει μια εργασία για επίλυση του προβλήματος. Διαφορετικά μπορεί να οδηγήσει σε κυρώσεις οικονομικού τύπου. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γίνονται σεβαστοί κοινοτικοί κανόνε. Και ο Επίτροπο ο κ. Σαβραμόπουλος στην Ολομέλεια είπε ότι θα επιβληθούν κυρώσει. Λοιπόν, ελπίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επιβάλλει το σεβασμό των συμφωνιών. Αυτή είναι η βούληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν είναι μια προσωπική θέση. Το Κοινοβούλιο ψήφισε ένα κείμενο σαφέστατο. Και στις ιτελικές εφημερίδες ε, δημοσιεύθηκε σαφέστατα το κείμενο και θέλουμε να εφαρμοστεί η αρχή της αλληλεγγύης. Ε, Είπατε πρόσφατα ήταν από του λίγου πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πήγε συνεδρίαση τη Επιτροπή των Περιφερειών τη Ευρώπη και διαβεβαίωσε ότι η μάχη για τη διατήρηση και μετά τον Brexit τη χρήση των ε, διαθωτικών τομείων θα διατηρηθεί με προσπάθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μαζί με την Επιτροπή των Περιφερειών. Τι γίνεται με τη γερμανική πρόταση όμω, παρέμβαση όσον αφορά τι οικονομικέ πικοδοτήσει των περιφερειακών ταμείων, που θα είναι ένα μέτρο που θα πλήξει τις χώρες εκείνες που δεν σέβονται τη συμφωνία για την ανακατανομή ε, των ε, μεταναστών. Απάντηση. Το κείμενο του Κοινοβουλίου αναφέρεται σε διάφορα μέτρα συμπεριλαμβανομένε κριτικασίας διαδικασία κατά παράβαση, που αυτή η διαδικασία οδηγεί και σε οικονομικέ κυρώσει. Εάν οι οικονομικέ κυρώσει επιβληθούν, είναι αδιάφορο πώ θα εφαρμοστούν η μέθοδος θα υποχρεωθεί ένα κάτω μέσο που συμμορφώνεται να πληρώσει λίγο πολύ ε, την αντιστοιχεία της ζημίας που προκαλεί στις άλλες. Ευχαριστώ όλους. Νομίζω ότι θα συνεχίσετε τώρα με τη συζήτηση ε, με τις παρεμβάσεις των εκπροσώπων των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Σας ευχαριστώ. Είστε πανίδιν, λέει ο κ. Σταγιάννη. Okay. Um, we, we... Λοιπόν, θα συνεχίσουμε τώρα με τα τελευταία 15 λεπτά για ερωτήσεις. Θα καλέσω λοιπόν τους εκπροσώπους των μη κυβερνητικών οργανώσεων να έρθουν εδώ και πρέπει πραγματικά να είμαστε πολύ σύντομοι γιατί η διερμηνία θα σταματήσει στις 12 και 4. Σας παρακαλώ λοιπόν να έρθετε, να καθίσετε για τα τελευταία 15 λεπτά. Okay. Uh, λοιπόν, ας ε, συνεχίσουμε. Συνεχίζουμε τη συζήτηση με τους προσκεκλημένους μας στο πάνελ. Ακούσαμε τους ομιλητές λοιπόν, ακούσαμε τις εμπειρίες τους, τις απόψεις τους για τη δουλειά τους, με τους ετούντες άσυλο, τους πρόσφυγες και τους μετανάστες σε διάφορα μέρη της Ευρώπης. Ας έχουμε τώρα ερωτήσεις παρακαλώ. Λοιπόν, ο κύριος εκεί και μετά εδώ η κυρία και η κυρία. Παρακαλώ. Μιχαλεύς από την ε, Τσεχία. Θέλω να ρωτήσω για το ζήτημα της Λετωνίας είπατε, είπε η κυρία Λάτσε, ότι ένα από τα προβλήματα είναι ότι υπάρχει ελάχιστη στήριξη στους πρόσφυγες. Οπότε, τι ποσό πιστεύετε εσείς ότι θα βοηθούσε να λυθεί αυτό το πρόβλημα, γιατί λέτε ότι παίρνουν πολύ λίγα. Πόσα θα έπρεπε να παίρνουν οι πρόσφυγες για να παραμείνουν στην Λετωνία. Και επίσης, Αναφερθήκατε και στο πρόβλημα εκμάθησης της γλώσσας. Αν τους επέτρεπαν η Λετωνία να μάθουν Ρώσικα, μήπως αυτό θα διευκόλυνε κάπως την κατάσταση. Απάντηση για το ποσό. Πριν ήταν 256 ευρώ και ήταν, είχε εκτιμηθεί πολύ χαμηλό το ποσό από την ΥΠΑΤΗ αρμοστή για τους πρόσφυγες στο ΙΕ. Το θέμα όμως δεν είναι ποιο θα πρέπει να είναι το ακριβές ποσό. Το θέμα είναι άλλου είδους στήριξη που χρειάζονται οι άνθρωποι αυτοί. Στέγαση, αν ε, τους προσφερθεί στέγαση, δεν πρέπει να αυξηθεί το ποσό. Επίσης, αυτοί που αναγνωρίζονται ως πρόσφυγες και ότι χρήζουν επικουρικής βοήθειας. Αυτοί χαίρουν άλλων πλέον εκτιμάτων εξαιτίας αυτού του καθεστώτος. Τώρα για τη ρύθμιση του γλωσσικού. Δεν νομίζω ότι το θέμα εδώ είναι να μάθω μια άλλη γλώσσα. Ίσως να γίνουν πιο ήπιες οι προϋποθέσεις για να βρει κανείς δουλειά. Αλλά πώς θα είναι σε επαφή με τους πελάτες, με τους ντόπιου. Δεν θα πρέπει να γνωρίζουν κάποια ελάχιστα λετονικά. Είναι δύσκολο βέβαια να πάει κανείς να παρακολουθήσει μαθήματα. Τρεις μήνες δεν φτάνουν. Οπότε ίσως θα πρέπει να γίνουν πιο επίσης συνθήκες, οι απαιτήσει και με το που φτάνουν να αρχίσουν να μαθαίνουν τη γλώσσα πιο εντατικά. Ευχαριστούμε. Και εσείς θέλετε να απαντήσετε σε αυτό, ε? Ναι. Και εγώ θέλω να αναφερθώ στην κοινωνική προστασία. Το επίπεδο πρέπει να είναι ίδιο για όλους. Το επίπεδο κοινωνικής προστασίας πρέπει να είναι το ίδιο για όλους. Τον υπάρχουν μηχανισμοί διάκρισης όσον αφορά την κοινωνική προστασία ανάμεσα στον τόπιο πληθυσμό και τους ετούντες άσυλο ή τους γνωρισμένους πρόσφυγες δεν λειτουργεί. Όταν προσπαθούμε να δούμε ποιο είναι το επίπεδο κοινωνικής προστασίας που χρειάζεται, πρέπει να λέμε υπόψη μας δύο στοιχεία. Το πρώτο είναι, είναι το όριο φτώχειας, για να υπάρχει κοινωνική προστασία για όλους και αυτός πρέπει να είναι ο βασικός κανόνας ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, για όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέμα που τίθεται όμω είναι οι άνθρωποι αυτοί μπορούν σε περιοχές κοινωνικής προστασίας να κατασταθούν μόνιμα και μπορούμε να στηρίξουμε αυτέ τι περιοχέ. Οπότε ποια είναι η δυνατότητα 56% των ανθρώπων που είναι πρόσφυγες στο Βέλγιο εργάζονται. Μετά από τέσσερα χρόνια λοιπόν συνεισφέρουν στην οικονομία. Οι οικονομικές μελέτες δείχνουν ότι οι πρόσφυγες συνεισφέρουν, καθαρή καθαροί στο ΑΕΠ των χωρών. Το ζήτημα λοιπόν είναι ποιο θα είναι το διάστημα της μεταβατικής περίοδου και πώς αυτό θα είναι όσο γίνεται πιο μικρό αυτοί που δουλεύουν για την απασχόληση των προσφύγων ή για τη δημιουργία οικονομικής δραστηριότητας ξέρουν τι πρέπει να γίνει. Να υπάρχουν μηχανισμοί που να βοηθούν εύκολα να περάσει κανείς από την κοινωνική προστασία στην ενεργό οικονομική δραστηριότητα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ευχαριστούμε. Επόμενη ερώτηση παρακαλώ. Εσείς. Η ερώτησή μου απευθύνεται σε όποιον θέλει να μου απαντήσει βλέπουμε ότι η προσπάθεια της Ευρώπης σήμερα είναι να σπάσει την προσπάθεια των προσφύγων να φτάνουν στην Ευρώπη. Είναι αυτό ιδανικό σε μια Ευρώπη που έχει τόσες πολλές διαφορές. Δηλαδή, καλά κάνουμε και ψάχνουμε κάτι τέτοιο. Ποιος θέλει να απαντήσει. Εγώ θα προσπαθήσω να απαντήσω. Αυτή η δευτερογενής μετακίνηση είναι κάτι το οποίο βλέπουμε στις βαλτικές χώρες. Έτσι κι αλλιώς δεν μπορούμε να υποχρώσουμε κανένα να μείνει στη χώρα μας. Αποκλείται να τα καταφέρουμε, εκτός να θέλουμε να κλείσουμε εντελώς τα σύνορα και να έχουμε ελέγχους και να τους υποχρώσουμε να μείνουμε. Αλλά δεν είναι αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε. Θέλουμε να μείνουμε στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προσφέρει ανθρώπινα δικαιώματα και εξωπρεπείς συνθήκες διαβίωσης. Δεν μπορούμε να τους υποχρώσουμε να μείνουν λοιπόν. Πρέπει να τους προσφέρουμε όμως ευκαιρίες για να μείνουν, να δημιουργήσουμε μια τέτοια κατάσταση. Το είπε και ο κύριος Φαντέρε νωρίτερα, ότι υπάρχει το σημείο εκκίνησης, ότι δηλαδή τους βοηθούμε να γίνουν ουσιαστικά μέλη της κοινωνίας. Αυτό που κάνουν πολλές χώρες όμως επίτηδες είναι να μην προσφέρουν τέτοιες ευκαιρίες και προωθούν αυτό το δευτερογενές ε, κίνημα, αυτή τη μετακίνηση την ε, δευτερογενή σε δεύτερο στάδιο. Άλλος κανείς που θέλει να απαντήσει σε αυτό. Ωραία. Λοιπόν, άλλος ποιος ήθελε να ρωτήσει κάτι. Εσείς. Οι δύο τελευταίες ερωτήσεις, εσείς οι δύο. Παρακαλώ. Γεια σας. Από την Ισπανία. Country, they all talk... Από την Ισπανία. Οι πρόσφυγες στη χώρα μου μιλάνε για κόλαση όταν φτάνουν ξανά από την αρχή, γραφειοκρατία ε, και λοιπά προβλήματα. Εσείς θα μπορούσατε να μου πείτε τη δική σας εμπειρία στην, ε, στον καθημερινό αγώνα. Θεωρείτε πως πρέπει να γίνει κάτι σε ευρωπαϊκό επίπεδο έτσι ώστε να τους βοηθήσουμε με αυτόν τον τρόπο. και η επόμενη ερώτηση και μετά θα ολοκληρώσουμε τις απαντήσεις. Στην κυρία Λάτσα θα ήθελα να απευθύνω μια ερώτηση. Αναφέρατε πως υπάρχουν κάποιες χώρες που προωθούν αυτές τις δευτερογενείς μετακινήσεις. Εννοείται πως και η Λετωνία είναι μία από αυτές τις χώρες που στηρίζει αυτές τις ε, μετακινήσεις. Δεν νομίζω πως αυτή είναι η πρόθεσή μας αλλά νομίζω πως ε, δεν μπορώ να πω κιόλα πως ε, δεν χαίρονται που φεύγουν οι πολιτικοί μας. Το σύστημά μας, είναι η αλήθεια, ε, δεν έχει ακόμα τη δυνατότητα να κάνει πολλά. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ήθελα λοιπόν να δώσω τώρα 30 δευτερόλεπτα στον καθένα από εσά για να ολοκληρώσει και ίσως να απαντήσει για το θέμα της γραφειοκρατίας. Γερμανία και γραφειοκρατία. Είναι κόλαση τα πράγματα, μπορείτε να το Φανταστείτε, σίγουρα δεν είναι καθόλου εύκολα τα πράγματα, ούτε για μα. Όταν κάποιο πρέπει να κάνει κάτι, πρέπει να συμπληρώσει ένα έντυπο. Για να συμπληρώσει ένα έντυπο, θε τρία άλλα έντυπα. Φανταστείτε πόσο αυξάνεται η γραφειοκρατία. Εμεί έχουμε κάποιε εταιρικέ σχέσει, έχουμε κάποιε συνεργασίε με το δημόσιο, μα στέλνουν κάποιου δημόσιου υπαλλήλου για να μα βοηθήσουν στη συμπλήρωση εντύπων. Αλλά εκεί που νομίζει ότι έχει καταλάβει τι γίνεται, Θέλει και άλλο. Χρειάζεται και άλλη γραφειοκρατία. Μετά, όταν υπάρχουν πολλέ μη κυβερνικέ οργανώσει που συνεργάζονται και πρέπει να ε, μεταφράσουν ένα έντυπο και εκεί υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχουν λοιπόν γενικότερα προβλήματα γραφειοκρατίας που καθυστερούν τα πράγματα. Και αυτά τα έντυπα πρέπει να συμπληρώσει κάποιος είναι βασικά πράγματα για να βρει ας πούμε διαμέρισμα. Δεν ξέρω τι γίνεται στις άλλες χώρες, αλλά η γραφειοκρατία στη Γερμανία είναι τερατώδης. Αν πάρω κι εγώ για το θέμα του άδειας διαμονής, ένα ζητά να αποκτήσει άδεια διαμονής, το γραφείο των ε, εξωτερικών αλλοδαπών αρνείται, οπότε κάνει προσφυγή το άτομο μετά στο Συμβούλιο Εφετών για τους Αλοδαπούς όταν η προσφυγή οδηγήσει στο, Συμβούλιο να ανατρέψει την απόφαση του Γραφείου Αλλοδαπών, αποσύρει την απόφαση του το Γραφείο Αλλοδαπών πριν την απόφαση της δικαιοσύνης και ξαναπαίρνει νέα απόφαση που εκ νέου είναι αρνητική και αυτό εμποδίζει το δικαστήριο να τοποθετηθεί επί της αποφάσεως. Και αυτό το γαϊτανάκι μπορεί να φτάσει μέχρι 9, 10, 11 φορές. Η πιο σοβαρή υπόθεση ήταν 11 φορές να γίνεται αυτό, διότι το δικαστήριο θα αποφάσιζε να ανατρέψει την απόφαση της υπηρεσίας αλλοδαπών, η υπηρεσία αλλοδαπών αποσύρει την απόφασή της. Καταλαβαίνετε το κόστος, το διοικητικό κόστος που εκπροσωπεί αυτό, αυτό το γαϊτανάκι που από πλευράς νομικής είναι σχεδικό, σχεδόν να πούμε κολυσιεργία και συνενοχή των δημοσίων υπαλλήλων. Είναι σοβαρό αυτό. Ο κύριος Κόβατς, ε, γρήγορα, ποια ήταν η εμπειρία μας ότι η γραφειοκρατία μπορεί να είναι προβληματική για τον κόσμο, αλλά ε, δεν είναι αυτή μόνο που σχετίζεται με το άσυλο και ε, ε τους πρόσφυγες η γραφειοκρατία στην Ουγγαρία είναι από τι πιο δύσκολε. γενικά για όλου. Αλλά όσον αφορά και τις χρόνες καταγωγή των ανθρώπων αυτών ε, και εκεί αντιμετωπίζεται η γραφειοκρατία. Αν είσαι από μια χώρα η οποία είναι σχεδόν ανύπαρκτη και πρέπει να ακολουθήσει γραφειοκρατικέ διαδικασίε, ίσω να είναι πάρα πολύ δύσκολα τα... Άμα δεν υπάρχουν εκεί διαδικασίε. δύσκολο να μάθει ότι υπάρχουν προθεσμίε και έντυπα να συμπληρώσεις και και διάφορε γραφειοκρατικέ διαδικασίε. Και αν έχει από μια χώρα όπου είναι διεφθαρμένη η γραφειοκρατία, μπορεί να βρει πολύ διαφανή την Ουγγρική γραφειοκρατία, πολύ ομαλή και πολύ εύκολη. Άρα ποικίλουν οι υποθέσει ανάλογα με το άτομο και πού προέρχεται. Το μόνο πρόβλημα που αφορά μόνο τους πρόσφυγες και που αντιμετωπίζεται που αφορα μονο του προσφυγε και που αντιμετωπιζεται είναι η άγνοια ε, ε των, ε, των του διοικητικού προσωπικού των διαφόρων θεσμικών οργάνων. Πρέπει να του ενημερώσουμε, α πούμε, ότι οι πρόσφυγε έχουν τα ίδια δικαιώματα όπω οι Ούγγροι πολίτε, ούτως ώστε να μην πρέπει να φοβούνται για την αποδοχή ε, αιτήσεων ε, και πρέπει ε, να ασχολούνται καθημερινά με τις υποθέσεις και πρέπει να ενημερώνουν τα άτομα που θα πρέπει να, είναι ενήμεροι υπάλληλοι παρά να κάνουν συστημική αλλαγή. Ορίστε. Λοιπόν, μια που άνοιξα εγώ την ε, συζήτηση, σε αυτό το πάνελ, ας μου δοθεί και η ευκαιρία να κλείσω τη συζήτηση. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή. Ε, πιστεύω, μετά από την ε, πείρα μου πάνω σε αυτό το θέμα που λέγεται φιλοξενία ε, και ό, που εμπεριέχει και το άσυλο και το, την, την, και το relocation, την επανένωση οικογενειών, θα πρέπει να υπάρξει ε, άμεση και σωστή ενημέρωση και πληροφόρηση των ανθρώπων που θέλουν να μετακινηθούν από τις χώρες τους για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν εκεί. Αυτό λοιπόν που δεν υπάρχει είναι η άμεση και η σωστή πληροφόρηση. Αυτό λοιπόν εξαρτάται από εσά. Εξαρτάται από τις εκάστοτε κυβερνήσεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πώς θα μπορέσουν να χτίσουν ένα καλό πυλώνα ενημέρωσης όλων αυτών. Από εκεί και πέρα είμαι σίγουρος ότι πολλά θέματα θα πάρουν ε, καλύτερη, καλύτερη μπορώ να πω θα υπάρξει καλύτερη έκβαση σε πολλά θέματα όπως είναι το άσυλο και το, η, επανασύνδεση οικογενειών. Καθημερινά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στο πεδίο είναι ερωτήσεις ασύλου, επανασύνδεσης και αβεβαιότητας. Αβεβαιότητας, ακούσαμε όλους τους συνομιλητές εδώ πέρα, ο καθένας ξεχωριστά από τις χώρες του, αβεβαιότητα το τι γίνεται στη Γερμανία, το τι γίνεται στην Ουγγαρία, το τι γίνεται στην Αυστρία, το τι γίνεται στη Γαλλία. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια κεντρική τράπεζα δεδομένων και πληροφοριών επιτέλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα λέει τα πράγματα με το όνομά του. Για να πάρει άσυλο πρέπει να είσαι έτσι, για να επανενωθεί με την οικογένεια σου θα πρέπει να κάνει αυτό και από εκεί και πέρα να κάτσουν όλε οι χώρε κάτω από αυτή την ομπρέλα κοινή πορεία στην ενημέρωση και στι πληροφορίε. Για μένα προσωπικά η πληροφορία είναι η αρχή του παντός. Και του καλού και του κακού. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Thank you very much. Um... Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ όλους που απαντήσατε σε ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και παρακολουθήσατε το σεμινάριο. Ευχαριστούμε πολύ και τους διερμηνείς. Έχω κάποιες ανακοινώσεις πρωτού τελειώσουμε. Οι φωτογραφίες, τα βίντεο και η ηχογράφηση όλου του σεμιναρίου θα σας σταλεί με email σήμερα το απόγευμα. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο είναι ελεύθερα για κατέβασμα, μπορείτε να τα αποθηκεύσετε, να τα μοιραστείτε, αλλά να σας ζητήσουμε να ε, μονάσετε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αν το κάνετε. Επίσης, στην ε, οπτικοακουστική υπηρεσία του Κοινοβουλίου υπάρχουν ε, τα βίντεο των ε, άλλων εργαστηρίων και όλοι θα λάβετε ένα link για μια έρευνα, μπορείτε να συμπληρώσετε διαδικτυακά γιατί θα θέλαμε την άποψή σα για το σεμινάριο και τις ιδέες σας για το τι θα θέλατε να δείτε στο μέλλον, τι σας άρεσε, τι σας άρεσε λιγότερο κτλ. Και να πω ότι όσοι δεν υπέγραψαν το παρουσιολόγιο θα βρείτε τη συνάδελφό μου την Άννα εκεί πίσω και μπορείτε να υπογράψετε φεύγοντα. Σα ευχαριστώ λοιπόν ξανά. Εδώ φτάσαμε στο τέλο του σεμιναρίου.